Καλημέρα ε, σε όλους. Θα προεδρεύσω στα Ισπανικά. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω όλους στα Ισπανικά. Καλημέρα σας. Τα πρώτα μου λόγια ως αντιπρόεδρος είναι λόγια ευχαριστίας. Παρόλο που είναι πάρα πολύ λίγοι βουλευτές παρόντες, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη χθεσινή μου εκλογή και πάμε αμέσω χωρί αναισθητικό με το καλημέρα σας, με την εκλογή μου, μου πέσε ο κλήρο. Είναι πολύ δύσκολο να αντικαθιστάς τον Παύλο Σάλβα που ήταν σπουδαίος αντιπρόεδρος, συντονιστής και πάρα πολύ καλός μου φίλος. Ε, και θα προσπαθήσω όχι να σας κάνω να το ξεχάσετε, αλλά ε, να τον αντικατεστήσω επάξια και να το θυμόμαστε με νοσταλγία. Λοιπόν, πάμε στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε το σημείο 8. Είναι αιτήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μετά την απόφαση της διάσκεψη των Προέδρων στι αρχές του έτους έχουμε μια νέα κατανομή αρμοδιοτήτων ε, ανάμεσα στον ετήσιο έλεγχο και Ε, της έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΚΟΝ. Θα δώσουμε αμέσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κίρτσο. Παρακαλώ, κύριε Κίρτσο, έχετε το λόγο. Thank you, So, have this report. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι ε, έχω καταρτήσει την εκθεσή μου και έχω δεχθεί περίπου 316 τροπολογίες. Η διαδικασία που θα ακολουθήσω... Is that on the 6th of ε, February we'll have a discussion... Uh, no, sorry. Ε, we have, we'll have a shadow... shadow... Θα έχουμε λοιπόν στις 7 Δεκεμβρίου συζήτηση με τους και ηγητές για να συζητήσουμε τις τροπολογίες και για να προσπαθήσουμε να τις κατηγοριοποιήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε ενδεχομένως και ελπίζω και όλες να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Και κατόπιν η έκθεση θα ψηφιστεί και πάλι ελπίζω από την Επιτροπή στις 6 Φεβρουαρίου. Και θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Πριν από αυτό, ο κύριος Χόια, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα έρθει στην Ολομέλεια και θα τοποθετηθεί στις ερωτήσεις μας. Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε και θέλω να κάνω κάποιες γενικής φύσεως παρατηρήσεις για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Όπως σας είπα, δεχτήκαμε πάρα πολλές τροπολογίες που ε, ασχολούνται όλες με το θέμα το φορολογικό, κυρίως με το θέμα των ενδιάμεσων φορέων και επίσης και με την ε, ε, επικείμενη φορολογία, μάλλον νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα φορολογίας Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι ένας αποτελεσματικό φορέας βεβαίως θα τους ε, ζητήσουμε να προχωρήσουν τουλάχιστον όσον αφορά τα φορολογική φύσεως θέματα. Υπάρχουν όμως και πρακτικά θέματα. Παραδείγματος χάρη δεν μπορούμε να τους ζητήσουμε να δεχτούν αιτήματα που δεν είναι νομικά αποδεκτά. Μπορούμε αν θέλω ενδεχομένως ε, πολιτικά να το ζητήσουμε αυτό, αλλά επειδή είναι περίπλοκο το θέμα δεν θα το δεχτούν. Κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη δεν θα πρέπει να τους επιβαρύνουμε ιδιαίτερα με αιτήματα τα οποία κατ' ουσίαν έχουν να κάνουν με φορολογικές αρχές. Πρέπει βέβαια να επιμείνουμε να εφαρμόζουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προδιαγραφές για την αποφυγή της φόρο αποφυγής και των φορολογικών παραδείσων και επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων περιμένει από τους πελάτες της και αυτοί να εφαρμόζουν αυτές τις προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί. Πρέπει επίσης να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να στηρίξει τις ε, πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την φοροαποφυγή, κυρίως ε, στο ε, πλαίσιο ενός πακέτου το οποίο δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2016. Μία άλλη κατηγορία τροπολογιών έχει να κάνει με το στρατηγικό επενδυτικό πρόγραμμα, το ΕΦΣΥ, Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σε αυτήν την έκθεση δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάζουμε όλα τα θέματα του ΕΦΣΥ γιατί υπάρχει και μια ειδική έκθεση για το ΕΦΣΥ. Οφείλουμε όμως να επιμείνουμε έτσι ώστε το πρόγραμμα ΕΦΣΥ των στρατηγικών επενδύσεων να εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο που θα προάγει την συνοχή και θα ενισχύει την γεωγραφική κατανομή. Ε, Έχω ζητήσει και στατιστικά δεδομένα σχετικά με το εψί για να μπορώ να καταλήξω σε ένα αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να σα πω ότι όλα αυτά είναι λιγάκι περίπλοκα με την έννοια ότι τα περισσότερα κονδύλια διοχετεύονται σε μεγάλες οικονομίες, σε προηγμένες χώρες, αλλά αν κάνει κανείς ε, την ανάλυση των κονδυλίων με βάση το ΑΕΠ θα διαπιστώσει ότι η κατανομή τελικά είναι πράγματι υπέρ των μικρότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκείνων που έχουν διαρθρωτικά προβλήματα. Άρα δηλαδή όλα αυτά είναι ανοιχτά για αναλύσεις, για πολιτικές ερμηνείς αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε μέσα από τροπολογίες και με τη δική μου έκθεση να ε, αναφέρει τις προκλήσεις που υπάρχουν, κυρίως όσον αφορά τους στόχους της συνοχής. Μία τρίτη κατηγορία τροπολογιών έχει σχέση με το θέμα της εποπτείας που μπορεί να ασκήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήδη λειτουργεί μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο λογοδοσίας λογοδοτεί έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε αιτήσια βάση υπάρχουν ήδη τρεις, τρεις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δραστηριότητες ε, της ΕΤΕΠ ε, μια έκθεση την οποία κατάρτισε η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θέσεων και Επιτροπή Προεπολογισμών Εκεί αναφέρεται ο έλεγχος των ε, χρηματοψηφιακών δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ. Αυτή ε, καταρτίστηκε από την Επιτροπή ελέγχων του προπλογισμού και η τελευταία έκθεση που καταρτίστηκε από την Οικονομικών, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και από την Επιτροπή Προπολογισμών. Τρεις λοιπόν εκθέσεις. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι όσον αφορά τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΠ, εγώ είμαι υπέρ του να δημοσιεύεται μία περίληψη αυτών των πρακτικών, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα συμβάλλει στη διαφάνεια. Και η τέταρτη κατηγορία ε, τροπολογιών που έχουν κατατεθεί αφορά στις ε, δραστηριότητες για την κλιματική αλλαγή. 20,7 δις ευρώ. Αυτή είναι η χρηματοδότηση για το 2015. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δώσει ποτέ η ΕΤΕΠ. Η στρατηγική για το κλίμα της τράπεζας ε, λέει ότι θα πρέπει να ε, ξεπερνάνε οι χρηματοδοτήσεις το 25% της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και κατά τα άλλα η χρηματοδότηση της ΕΤΕΠ για τη νέα ενέργεια το 2015 ανήλθε σε 3,4 δις ευρώ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μία μείωση σε σχέση με το 2014, όπου το σχετικό ποσό ήταν 5,9 δις. Άρα δηλαδή υπάρχουν κάποια θέματα με την ε, κλιματική αλλαγή, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βρίσκεται σε σωστό δρόμο. Η πέμπτη κατηγορία τροπολογιών έχει σχέση με το θέμα των ε, προσφύγων και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Ε, υπάρχει πρόβλεψη υπέρ των χωρών τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, το προσφυγικό. Άρα δηλαδή και εκεί οφείλουμε να αναζητήσουμε τη δυνατότητα συμβαστικών προτάσεων, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα του προσφυγικού. Και τέλος ε, υπάρχει ένα έτσι, περίεργο θέμα, δεν θα μπω εδώ σε λεπτομέρειες για να σας το εξηγήσω, αλλά επειδή θα μπορούσε να είναι μια παγίδα, θέλω να πω ότι πολλές τροπολογίες έχουν σχέση με λεπτομέρειες που αφορούν σε μεμονωμένα προγράμματα. Άρα δηλαδή πρέπει να μελετήσουμε αυτά τα μεμονωμένα προγράμματα και καλείται η ΕΤΕΠ να δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα. Σε γενικές γραμμές, εγώ στον βαθμό τουλάχιστον του δυνατού θα ήθελα να αποφύγω να αρχίσουμε να εξετάζουμε συγκεκριμένα προγράμματα, δηλαδή να μπούμε σε λεπτομέρειες για θέματα που κατ' ουσίαν δεν γνωρίζουμε. Αυτή είναι η γενική εικόνα που σας και αγράφησα και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να καταλήξουμε στις ε, απαραίτητες λύσεις και συμβιβασμούς και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταθέσουμε μια ενδιαφέρουσα έκθεση η οποία θα ικανοποιήσει τουλάχιστον τους περισσότερους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κίρτσον. Σκιώδης τώρα. Από τους Η κυρία Μπερές, αντικαθιστά το σκιώδη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε στα νέα σας καθήκοντα. Και εγώ λέγομαι τώρα κύριο Ιβάν Καταλήν. Ζητώ συγγνώμη ε, ονόματος και εισηγητού, γιατί έχουν ε, ε, προεκλογικό αγώνα στη Ρουμανία και δεν είχε ληφθεί υπόψη αυτό όταν εγγράφηκε στην μέση διάταξη ακυρώθηκαν οι συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών. Ελπίζω να ξαναρχίσουν την άλλη εβδομάδα. Θα πρέπει ε, να δούμε τους συμβιβασμού και να διευκρινίσουμε. Πριν πω στην ουσία του κειμένου, σημειώνω ότι η τελευταία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για να το πω έτσι ευγενικά, δεν μας ικανοποίησε πλήρως. Μα λέει ο εισηγητή ότι ο κύριο Χόιερ θα έρθει στην Ολομέλεια. Μπράβο του, πολύ ωραία θα κάνει. Αλλά ε, μήπω να πούμε στον κύριο Χόιερ ότι δεν απαγορεύεται όταν συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έρχεται και στην ΕΚΟΝ καμιά φορά ε, και θα μπορούσε να απαντήσει σε ανησυχίε των βουλευτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση αυτή τη δομή. Πολύ δε περισσότερο που εκπρόσωπό του όταν ήρθε, πώς να το πω, είχε το θράσος, ε, όχι ακριβώς να υβρίσει, αλλά να επικρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δεν ε, ε, ήταν πάντα προσοχή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να υπογράφει τα διάφορα πράγματα που γίνονται ερήμην του. Κάποια πράγματα λοιπόν εκεί πρέπει να διορθωθούν. Θα έλεγα κατά τον ίδιο τρόπο ότι υπάρχουν δύο-τρία θέματα πάρα πολύ κρίσιμα, τα ανέφερε και ο εισηγητής, ίσως να σας το φωτίσω από μια άλλη σκοπιά. Το πρώτο, ίσως μια γενική παρατήρηση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα πρέπει να είναι υποδειγματική. Είναι η μεγάλη ενιαία Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Θα πρέπει να είναι υποδειγματική και ας προς τη διακυβέρνησή της και ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά τα φορολογικά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μπορεί να εθελοτυφλεί ή να ε, αμελεί ε, κάποιες φορολογικές ε, συμπεριφορές των εταίρων της, είτε είναι κράτη είτε είναι επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να είναι φορέας χρηστής διακυβέρνησης με την αυστηρή και κυριολεκτική έννοια και για τον εαυτό της και για τους εταίρους της. Και από ό,τι φαίνεται, πέρα από τα ωραία λόγια εκεί, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά να γίνουν και να ελεγχθούν. Ελπίζω ε, η έκθεση αυτή ε, να βοηθήσει να προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή, είπε ο συγητής ότι ήταν ε, πάρα πολύ περίπλοκο, τα στοιχεία ήταν πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, ποιο είναι το πνεύμα κατά την άποψή μου της επέμβασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνη, ένα στίχημα βάλαμε Ενδεχόμενοι εμείς ε, να αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ΕΤΕΠ ε, την εφαρμογή του σχεδίου στρατηγικών επενδύσεων του Juncker, να είναι εργαλείο δηλαδή για να προχωρήσει η διακυβέρνηση και οι βέλτιστες πρακτικές. Βεβαίω, τράπεζα είναι, κέρδη θέλει να έχει και να είναι και κερδοφόρα γενικά ως ίδρυμα, αλλά θα πρέπει να φροντίσει να υπάρχει μια γεωγραφική εξισορρόπηση και να ε, υποστηρίζει τις δημόσιες επενδύσεις εκεί που ε, οι ιδιώτες δεν έρχονται να επενδύσουν ε, έτσι, φυσικά. Δύο τελευταία σχόλια. Πρώτον, για την εφαρμογή των συμπερασμάτων των συμφωνιών του Περισιού Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία μιας στρατηγικής για την μετάβαση, την οικολογική και χαίρομαι που κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Συμβούλιο ετέθη αυτό. Εμείς είχαμε ζητήσει στο σχέδιο Juncker 1 κάποια πράγματα τα οποία θα περάσουν στο δεύτερο ε, σχέδιο Juncker. Να υπάρχει ειδική μέρημνα και μνήμα γι' αυτά. Και τέλος κύριε Σιγητά θα πρέπει να δούμε τι επίπτωση θα έχει το Brexit ε, στη λειτουργία της ΕΤΕΠ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη στρατηγική επενδύσεων. Ζητώ συγγνώμη πρόεδρε, μακρηγόρησα πάρα πολύ. Και δεν με κόψατε. Εντάξει, πρώτη φορά προεδρεύω, θα μάθω. Ε, muchas gracias. Ahora, en nombre de, de ECR... Ε, από την ECR, ποιος θέλει το λόγο, κανείς. Ε, la señora López Bermejo tiene la palabra. Buenos días y gracias, presidente. Η κυρία Λόπες Μπερμέχο. Ε, ε, το θέμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ε, πρέπει να πω ότι ο κόσμος δεν τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ούτε το σχέδιο Juncker ούτε την Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, και κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια προβλήματα. Η ΕΤΕΠ δεν έχει ούτε τις διοικητικές δομές ούτε την πολιτική βούληση έτσι ώστε να πάνε στις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, οι πιστώσεις και τα δάνεια και στην πραγματική οικονομία. Είμαστε ε, πραγματικά ε, δέσμοι των πάρα πολύ μεγάλων έργων ε, που είναι κερδοσκοπικά και δεν βοηθούν την κοινωνία στην οποία υλοποιούνται. Υπάρχει και ένας συντηρητισμός λένε ορισμένοι. Εγώ θα το έλεγα διαπλοκή ε, και συνενοχή ε, με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και χρηματοπιστωτικά. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, προφανές στο πώς συνδέεται η ΕΤΕΠ με τις δημόσιες αρχές και την κοινωνία των πολιτών. Είναι μια καχυποψία αυτή που διέπει τη σχέση τους και τους θεωρεί πολλές φορές εμπόδια στην ιδιωτικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, είναι σε θέση να φέρει δημόσια κονδύλια σε εκείνους που τα χρειάζονται και πρέπει να είναι η σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας για την περιφερειακή συνοχή, την κοινωνική συνοχή. Μια τελευταία ε, υπόθεση. Είναι ε, πάρα πολύ αδιαφανής η διαχείριση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, καταγγέλουμε ε, τη δράση της στην Παλαιστίνη, στα κατεχόμενα συγκεκριμένα. Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία έχουμε καταγγείλει στην COP22 σε σχέση με τη Δυτική Σαχάρα. Υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει ο χάρτης των θεμελιδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ε, δεσμεύεται και η ΕΤΕΠ από αυτή διότι διέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες γενικά. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή προς μια πιο δημοκρατική και χρήσιμη ΕΤΕΠ για τον ευρωπαϊκό λαό αλλά και τους γείτονε λαούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λόπες Μπερμέχο. Από τους Πρασίνους, ο κύριος ε, Λάμπερς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Κίτσο, σας άκουσα προσεκτικότατα και ξέρετε κάποιε φορές αναρωτιέμαι, εάν εδώ συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει εκτό αυτής της αίθουσα, εκτό του κοινοβουλίου. Διότι όταν σα ακούω να λέτε όλα πάνε καλά, η ΕΤΕ κάνει τη δουλειά τη, σέβεται τη θητεία τη και την εντολή τη. Ναι, κάποιε χώρε πρέπει να κάνουν περισσότερα, αλλά οι χώρε αυτέ τελικά παίρνουν το δίκαιο μερίδιό του, κάποιε έχουν αρκετέ επενδύσει κτλ. Μπορεί δηλαδή κανεί να πει ότι βάσει των κανόνων όλα πάνε καλά. Και ο Κρήτον το έλεγε αυτό. Αλλά αν κοιτάξουμε τι ισχύει στα χαρτιά, όλα μπορεί να πηγαίνουν καλά. Πώ θα πείσουμε όμω του υπόλοιπου. Εδώ να υπογραμμίσω δύο-τρία πράγματα που θα τα βάλω και σε τροπολογίε. Για να δείξω ότι κατά την άποψή μου δεν πάνε όλα καλά, για να μην πω ότι όλα πάνε πολύ στραβά. Και αν δεν το πούμε εμεί στο κοινοβούλιο, ποιο θα το πει αυτό. Να ξεκινήσω λέγοντα το 90%. 90% των επενδύσεων του ε, στρατηγικού ταμείου πηγαίνουν στου 15 τη Ένωση. και τα μισά πηγαίνουν στι μεγάλε χώρε. Μπορείτε να μου πείτε, ε, ωραία, μπορείτε να μα λέτε ότι η Γερμανία παίρνει το δίκαιο μερίδιο τη. Όμω το δίκαιο μερίδιο τη ε, Γερμανία ε, δεν θα έπρεπε να είναι μηδέν. Η χώρα αυτή έχει πραγματικά υπερβολική ρευστότητα, έχει πολύ χρήμα. Η Γερμανία θα έπρεπε να επενδύει πολύ περισσότερο και δεν το κάνει. Γιατί, γιατί το έψη η ΕΤΕ να χαλάνε έστω και μια δεκάρα, ένα λεπτό του ευρώ στη χώρα αυτή. Οι επενδυτικέ του δυνατότητε είναι μια πραγματικότητα. Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία παίρνουν λιγότερο ή περισσότερο από το δίκαιο μερίδιο του θα πει τίποτα. Όλη η προσπάθεια θα πρέπει να πηγαίνει στι περιοχέ όπου οι επενδύσει είναι απαραίτητε. Όπου οι επενδύσει και οι δυνατότητε δεν υπάρχουν. Δεύτερον, όταν μιλάμε με επενδυτικέ τράπεζε, τι μα λένε. Ότι η ΕΤΕ διαρκώ θα έπρεπε να αναλαμβάνει τα επικίνδυνα τμήματα, αλλά να αναλαμβάνει τα ασφαλέστερα των επενδύσεων. Και η ΕΤΕ σχεδιάζει προγράμματα που ο καθένα θα μπορούσε έτσι κι αλλιώ να προσθέσει. Η προσθετικότητα λοιπόν δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάλυψη του κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν να ε, ζητήσουμε από την ΕΤΕ να αναλάβει εδώ την ε, ε ηγεσία, όχι να μην είναι ουραγό. Πού είναι το δίκαιο μερίδιο ανάληψη κινδύνου. Δεν υπάρχει καμία, κανένα σχετικό ρόλο. Και αν δείτε και το χρονοδιάγραμμα, έχουμε φτάσει στα μισά του πρώτου βήματο, ε, τη πρώτη φάση του ΕΦΣΙ τέλο πάντων και μόνο 33% των επενδύσεων έχουν εγκριθεί και 20% έχουν υπογραφεί, έργα έχουν υπογραφεί. Άρα, ακόμη και αν χρειαστεί λίγος χρόνος για την επιτάχυνση και πάλι δεν είναι θερητικά αυτά τα δείγματα. Επίσης, ως προς την φύση των επενδύσεων, συνειδητοποιείται βεβαίως η ΕΤΕ το 25% των στόχων στις ανανεώσιμες το καλύπτει. Αν δείτε όμως τις τάσεις, τι φαίνεται. Οι επενδύσει στι ανανεώσιμε μειώνονται και μάλιστα πολύ έντονα, 20% πέρσι. Και οι επενδύσεις στα ορυκτά αναβαίνουν συν 25% των στόχων, αλλά ε, στα ορυκτά μάλλον συν 25%, μείον 25% στις ανανεώσιμες πηγές. Σε ποιον αιώνα βρισκόμαστε, είμαστε στην Ήπειρο Ευρώπη τον 21ο αιώνα, αυτό θέλαμε δεν συμβαίνουν αυτά που θελήσαμε. Η ΕΤ έκανε τα ανάποδα από αυτά που είχαμε ζητήσει. Ναι, μπορείτε να μου πείτε ότι εντάξει, στου πολιτικού ευθύνοντε μπορεί να ανταποκρίνονται σωστά, αλλά ε, πρέπει να ζητήσουμε από αυτού του πολιτικού ευθύνοντε, τον Κατάιναν πρώτον, να κάνουν αυτά που περιμέναμε. Γιατί επιτέλου η ε, ΕΤΕ χρηματοδοτεί προγράμματα και έργα του 19ου αιώνα. Θα έπρεπε να, να χρηματοδοτεί προγράμματα που να επιτρέπουν την ενεργειακή μετάβαση. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά αυτή θα είναι η φύση των τροπολογιών μα. Και πάλι, εάν αυτό το κοινοβούλιο δεν ακολουθεί μια νομικήστικη προσέγγιση, αλλά μια προσέγγιση τη ε, κοινή λογική και κοιτάξει τι πρέπει να γίνει, ε, εάν δεν το κάνουμε εμεί αυτό, ποιο θα το κάνει. Πρέπει να έχουμε και μια επαφή με την πραγματικότητα. Διότι πολλοί από εμά ε, περνάνε στα πολιτικά πράγματα ε, απομονωμένοι και αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάλλη από την ομάδα του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε αρμονικά για την έκθεσή του και ότι θα μπορέσουμε κάποιες από τις δικέ μας τις παρατηρήσει να τις ενσωματώσουμε. Διότι και τα τελευταία χρόνια κι εμείς έχουμε εργαστεί για τα θέματα αυτά με αφορμή τις προηγούμενες εκθέσεις. Θέλουμε λοιπόν απλώ να γίνει πληρέστερη έκθεση με ενδείξεις που έχουμε και από άλλες δουλειές, άλλες, από εκθέσεις σε άλλες επιτροπές που έχουν γίνει. Κάποια θέματα θεμελιώδου σημασία που μπορεί να έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, την διακυβέρνηση και την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Θα φροντίσω να τα υποβάλω σε τροπολογίε για να συνδυαστούν και με όσα κάνουν οι επιτροπέ τάξη και πάνω. Τώρα, αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχουν εργαλεία διακυβέρνησης και διαχείρισης για την αξιοπιστία των, ε, ε, των ενδιαμέσων και να δούμε τα προβλήματα διαφάνειας που μπορεί να υπάρχουν στην ΕΤΕ. Υπάρχουν αμφιλεγόμενα ζητήματα, ιδίως από την πλευρά των ε, οικονομικών ε, μεσαζόντων και με κατάληξη πολλές φορές φορολογικούς παραδείσους λέγεται εδώ λοιπόν δεν δίνει ποτέ τα λεπτομερή στοιχεία, τα λεπτομερή οικονομικά στοιχεία της ΕΤΕ η, των έργων μάλλον, των ε, επενδύσεων η ΕΤΕ ούτε τα δημόσια στοιχεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για του δημόσιου διαγωνισμού, τι δημόσιε προμήθειε που διοργανώνονται και επηρεάζει πολύ. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμεί ω Ιταλία το γνωρίζουμε πολύ καλά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και τη μαφία. Η υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να μην τα γνωρίζει τόσο, αλλά είναι σημαντικά για μα. Και επίση και κάποιε επικριτικέ παρατηρήσει για τα έργα τη ΕΤΕ ιδίως για τις επενδύσεις ε, σε υποδομές και τα σχετικά έργα. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Αυτά τα έργα θα πρέπει να έχουν και οικονομική κερδοφορία αλλά και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να έχουν και κοινωνικό, οικονομικό όφελος. Τα έργα αυτά δεν θα πρέπει να αφορούν απερχαιωμένες υποδομές ή επιλογές που μπορεί να θεωρηθούν μη ορθέ ανάλογα με τι τάσει τη αγορά. Λόγω χάρη αυτοκινητόδρομοι, οι οποίοι γίνονται με καταπροσέγγιση εκτιμήσει αρχικά και μετά βλέπουμε ότι η κυκλοφορία των ε, οχημάτων και των εμπορευμάτων τελικά δεν αυξάνεται, μειώνεται για λόγους που μπορεί να έχουν να κάνουν και με την ενεργειακή μετάβαση και το καθεξής. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποφύγουμε οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι να χρηματοδοτούν έργα και εγγυήσεις τέτοιου είδους. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει ο σχεδιασμός έργων και η υλοποίηση έργων με περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελο. Επίση και οι ιδιώτε εταίροι θα πρέπει να μπλέκονται στον όλο διάλογό μα, γιατί έχουμε εντοπίσει υποθέσει με αφορμή προηγούμενε εκθέσει, όπως αυτό που έγινε στο Μέστρε ή στην ε, Ισπανία λόγου χάρη, οι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση δεν ε, είχαν μπορέσει να έχουν εμπλοκή στην λοιπόν, του έργο και υπήρχαν ε, απώλειες για το δημόσιο σκέλος των δημόσιων οικονομικών. Εδώ λοιπόν θέλουμε υποδομές από την περιβαλλοντική οπτική γωνία να έχουν ένα καλό αντίκτυπο για τα δηληστήρια, για την αποθηκευσή άνθρακα, για τους αυτοκινητοδρόμους. Βλέπουμε να υπάρχουν κάποιο τέτοιου είδους ε, τα διαθέσεις από την πλευρά του προγράμματος Juncker, όμως ο Juncker και η Επιτροπή του στην πραγματικότητα δεν τα έχουν προωθήσει αυτά. Και δεν βλέπω γιατί το ταμείο αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο υποστήριξη εφόσον δεν πηγαίνει στην κατεύθυνση που θέλουμε δεν έχει καταφέρει το Στατικό Ταμείο να προσφέρει αυτή την ε, προστιθέμενη αξία στα έργα που θέλαμε και βασίζεται σε έργα τα οποία κατά την άποψή μας δεν είναι βιώσιμα από πλευρά περιβαλλοντική και κοινωνική. Και για την ενεργειακή μετάβαση, την ενεργειακή ανανέωση, ό,τι προβλέπετε περικόπτεται από, άλλα, από άλλες ε, επενδύσεις της ΕΤΕ. Λείπει λοιπόν η πρόβλεψη για την ανανέωση και την ανάπτυξη. Ελπίζω ο συγγητή να μπορέσει να σηματώσει κάποιε από τι παρατηρήσει μα στο κείμενό του για να υπάρχει και μια ευρύτερη απήχηση των απόψεων των υπόλοιπων ομάδων του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανεί άλλο το λόγο. Ε, από του κοιόδη συγγητέ, άλλο συνάδελφο, πριν ξαναδώσουμε το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Κανεί. Παρακαλώ, κύριε Κίρτσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε σε πολύ ενδιαφέρουσες συμβαστικές προτάσεις. Βεβαίως και θα επιθυμούσα και εγώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να είναι υποδειγματική τράπεζα, όπως είπε και η κυρία Περβάνς. Ε, Περές. Θεωρώ ότι ε, πράγματι μπορούμε να βελτιώσουμε τη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων. Υπάρχουν όμως ε, πρακτικές ε, δυσκολίες. Παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε, εγώ που έρχομαι από την Ελλάδα, πρέπει να σας πω, δεν έχουμε πλέον εθνική αναπτυξιακή τράπεζα και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Η ΕΤΕΠ ε, προσφέρει ένα τμήμα της ε, χρηματοδότησης. Αν δηλαδή το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι σε θέση να καλύψει το ποσοστό του που το αναλογεί στη χρηματοδότηση, τότε δεν μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και με αυτά, επ' αυτών, έχω συζητήσει και με την ΕΤΕΠ και με Έλληνες ε, οικονομολόγους, γιατί ξέρετε ότι η δική μου χώρα αντιμετωπίζει τα χειρότερα προβλήματα, διαρθρωτικά προβλήματα στην οικονομία μας ε, και είμαστε, χρειαζόμαστε πραγματικά επιγόντως επενδύσεις και υποστήριξη. Εμείς ε, στηρίζουμε τη Συμφωνία του Παρισιού και είμαι πεπισμένο ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε, κυρίως τώρα που θα ακολουθήσει η περίοδος ε, Τραμπ στις Ηνωμένε Πολιτείε. Επίσης, συμφωνώ ότι οφείλουμε να δούμε τι θα σημαίνει το Brexit, η έξοδος τη μεγάλη Βρετανίας για την ε, εξέλιξη της ΕΤΕΠ. Πάντως, ε, ξέρετε κάτι, θα επανέλθω με πιο ενδιαφέρουσα ανάλυση, αλλά πιστεύω ότι γενικά η ΕΤΕΠ ε, τίνει χείρα βοηθεία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι όλα τέλεια. Σωστό αυτό που ελέγχθη. Όμως, ανταυτού, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί στην κριτική μας. Γιατί σε τελική ανάλυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε πράγματα που είναι πολύ χειρότερα από το πώς λειτουργεί η ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρόλο που το είπε ο ε, επαναλαμβάνω το χρονοδιάγραμμα. 316 τροπολογίες έχει λήξει η προθεσμία, θα ψηφιστεί στις 6 Φεβρουαρίου για να πάει στην Ολομέλεια το Μάρτιο. 6 Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα 5 λεπτών μέχρι να έρθει ο κύριος Δάισελμπλουμ. Οικονομικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Eurogroup είναι το επόμενο θέμα μας. 5 λεπτά διάλειμμα.

So dear colleagues, good morning. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Καλωσορίζουμε τον Γερούν Ντάισελμπλουμ από την ιδιότητά του, του Προέδρου του Eurogroup της Ευρωομάδας για την ανταλλαγή απόψεων και τον οικονομικό διάλογο που έχουμε ως προς την εφαρμογή των συστάσεων ε, αναχώρα και το πρόσφατο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δέσμη μέτρου για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Γνωρίζουμε ότι την άλλη εβδομάδα έχει πολύ σημαντική συνεδρίαση το Eurogroup για τα θέματα αυτά και βεβαίως για κάποια άλλα θέματα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για τη δική μας Επιτροπή συμπεριλαμβανομένης και της περίφημης ε, ε, ε, σύστασης για την Ευρωζώνη. Ξέρω ότι διήστανται οι ε, απόψεις, αλλά κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ε, κοινή ε, φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο ε, του ενεργειακού, μάλλον του, του οικονομικού μείγματος που δεν μπορεί να επαφείται μόνο στα νομισματικά. Είναι και το θέμα ε, της Ελλάδας. Ε, γίνεται συζήτηση για τη δεύτερη αξιολόγηση αλλά και για τα μέτρα σχετικά με το χρέος. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και προσβλέπουμε σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Έχετε μέσα στο λόγο για την εισαγωγική σας ομιλία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμοι μέλη. Με χαρά έρχομαι στην Επιτροπή σας και πάλι για τον οικονομικό μας διάλογο. Στην παρέμβαση μου θα πω δύο λόγια για την οικονομική κατάσταση, για τα θέματα που έχουν απασχολήσει τους τελευταίους μήνες στην Ευρωομάδα, καθώς επίσης και τις προκλήσεις που μας περιμένουν, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας κύριε Πρόεδρε. Ε, οι προβλέψει για το φθινόπωρο του 2016 Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια ε, μετριοπαθής ε, ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι ε, η τέταρτη συνεχής χρονιά και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Αυξάνεται και η ανάπτυξη και το πραγματικό εισόδημα και η ιδιωτική ε, κατανάλωση. Θετικές εξέλιξεις. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε. Ε, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Παρά το γεγονός ότι ε, για κάποιο ε, καιρό μειώνεται, η ενεργεία παραμένει πάρα πολύ υψηλή σε κάποια μέρη της Ευρωζώνης. Επιπλέον, είχαμε ούριους ε, ανεμούς ε, παραδικά που έχουν αρχίσει τώρα να μειώνονται και αυξάνεται η αστάθεια και βεβαιότητα. Για την Ευρωζώνη τι σημαίνει αυτό. Τώρα περισσότερο από ποτέ έχει έρθει η ώρα να βεβαιωθούμε ότι η ανάκαμψή μας θα είναι πιο ε, και ποιο μπορεί να αυτό υποστηρίζεται. Αυτό χρειάζεται υγιή, ε, δημοσιονομική πολιτική, ε, διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές. Τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλο συμφέρον να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως ε, η συγκέντρωση μπορεί να είναι ε, η απάντηση για κάποια θέματα και αυτό αφορά ας πούμε, την Τραπεζική Ένωση, αλλά δεν είναι για όλα τα προβλήματα. Ταυτόχρονα χρειάζεται ένα συντονισμό στην Ευρωζώνη έτσι ώστε να ελεγχιστοποιήσουμε ε, τις ανητικές επιπτώσεις και να μεγιστοποιήσουμε τις θετικές επιπτώσεις και την μετάδοση σε άλλες χώρες. Αυτό κάνουμε για τις συζητήσεις μας θεματικές για την ανάπτυξη και τις θέσει εργασία. Μετά τις συστάσεις που έχουμε απευθύνει στην Ευρωζώνη και τα κράτη-μέλη και στόχος είναι να ενταθούν οι προσπάθειες μεταρρυθμιστικές με συνειδητοποίηση και ανταλλαγή απόψεων για διάφορους τομείς πολιτικής για το μέλλον. Ε, σκοπεύω να ενισχύσω την πίεση των ομοτήμων ε, για τις βέλτιστες πρακτικές, για την σύγκριση ε, μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα συνταξιωτικά συστήματα, τα βιώσιμα και το πλαίσιο για την αφαιρεγκαιότητα και τις πτωχεύσεις. Η ε, ανάπτυξη και η μεγέθυνση θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, έτσι ώστε οι πάντες να εποφελούνται από την ανάκαψη αυτή. Έρχομαι τώρα στο θέμα των φορολογικών πολιτικών των δημοσιονομικών πολιτικών. Ε, οι προσπάθειες εξυγίανσης των κρατών μελών αποδίδουν καρπούς. Η Eurostat ε, τον περασμένο μήνα δημοσίευσε τα στοιχεία ε, σε επίπεδο ευρώ. Στην ευρωζώνη είναι 2,1% γενικά το έλλειμμα σε σύγκριση με 6,2% που ήταν πριν από 6 χρόνια και αναμένεται να πέσει στο 1,8% κατά τη διάρκεια του 2016. Επίσης, το δημόσιο χρέος άρχισε να μειώνεται συνολικά στην Ευρωζώνη και έχει φτάσει στο 90,4%. Και οι προβλέψεις για το φθινόπωρο αναμένουν ε, τάση συνεχώς φθήνουσα. Ωστόσο, αυτό είναι μέση όρη και ε, κρύβουν κάποια ετερογένεια ε, και χρειάζεται να γίνει πρόοδος σε πολλά κράτη-μέλη έτσι ώστε να ενισχυθεί και να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και να μπορούν να απορροφούν τους κραδασμούς. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, εφαρμόζονται σωστά και με συνέπεια ε, τα ε, θέματα του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Θα ασχοληθεί το Eurogroup με τους προπολογισμούς των κρατών μελών στις 5 Δεκεμβρίου σε τακτική του συνεδρίαση. Σημείωσα τη συστάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζητεί επέκταση ε, μισή ε, εκατοστιαία μονάδα στις χώρες του ευρώ. Να σας πω δύο λόγια σχετικά. Ε, για να έχουμε από κοινού αξιοπιστία θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στα όσα λέμε και πράττουμε. Στη στάση αναχώρα έχουμε κάποιες συστάσεις που βασίζονται ε, στο Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Θα έχουμε συμφωνήσει ε, κατά τη διάρκεια του έτου και αυτά θα πρέπει να βρίσκουν ε, αντανάκλαση στο σχέδιο προπολογισμού των κρατών για το 2017. Ωστόσο αυτό θα ήταν διαφορετικό από την δημοσιονομική επέκταση που προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο, θα πρέπει να σεβόμαστε τα θεσμικά και τις ευθύνες μας. Δηλαδή, Όλοι οι προϋπολογισμοί θα πρέπει σταδιακά να έχουν ε, ο στόχο να είναι ισοσκελισμένοι. Ε, τώρα, ε, τα φορολογικά κίνητρα, μάλλον τα δημοσιονομικά κίνητρα είναι το θέμα. Θα πρέπει να εθαρρύνονται οι υπολογισμοί να δαπανούν περισσότερα. Σε κάποιες χώρες, ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την εντολή να κάνει συστάσεις για τα δημοσιονομικά, αλλά οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές να ε, εναπόκειται στις χώρες τις ίδιες να δουν πώς θα το αξιοποιήσουν αυτό. Το επόμενο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι η Τραπεζική Ένωση. Έχουν γίνει σημαντικές προοδοί τα τελευταία χρόνια. Ε, ε, το SRB έχει αρχίσει να λειτουργεί πλήρως και ο μηχανισμός, ο μηχανισμός εποπτείας SSM για την επόμενη διετία. Όλα τα κράτη-μέλη ε, έχουν μεταφέρει την οδηγία BRRD ε, για το θέμα της εξυγίασης ε, των τραπεζών και έχουν επίσης κυρώσει τη διακυβερνητική συμφωνία για το SRF. Όλες οι συμμετέχουσες χώρες σχεδόν έχουν υπογράψει εκτός από τέσσερις και προσπαθούμε να τις φέρουμε σε αυτό το δρόμο. Αυτό προετοίμασε το δρόμο έτσι ώστε να αρχίσει η τεχνική δουλειά ε, για το Single Resolution Fund, ε, ένα από τα στοιχεία που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Παραμένω πεπισμένο ότι μια καλώς λειτουργούσα τραπεζική ένωση είναι προαπαιτούμενο έτσι ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα η νομισματική ένωση. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις για την ενίσχυση τη ΟΝΕ. Πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ένωση τραπεζική και των κεφαλαίων αγορών. Ε, ένα σύστημα εγγύηση των καταθέσεων ε, θα βοηθήσει, χρειάζεται ίσους κανόνες ε, το παιχνίδι για να λειτουργήσει καλά. Και θα πρέπει οι συνομοθέτες γρήγορα να δώσουν συνέχεια στη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά. Τέλος θα ήθελα να πω δύο λόγια για την κατάσταση ε, των πραγμάτων σε σχέση με την Ελλάδα. Από τότε που είχαμε εδώ τον οικονομικό μας διάλογο, το Φεβρουάριο, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος ε, οι ε, ελληνικές αρχές, οι θεσμοί και το Eurobro κατάφεραν να κλείσουν την πρώτη αξιολόγηση. Η Ελλάδα έχει εφαρμόσει εντυπωσιακό κατάλογο μεταρρυθμίσεων ε, με βάση το πρόγραμμα που είχαμε συμφωνήσει αμοιβαία πέρυσι. Στις 24 Μαΐου στο Eurogroup καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία πλαίσιο, θα τη χαρακτηρίζα, για ε, μέτρα ενδεχόμενα για τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό συμπεριλαμβάνει βράχη πρόθεσμα μέτρα που έχει τελειώσει σε τεχνική βάση η εργασία αυτή και μέχρι το τέλος του προγράμματος, στα μέσα του 2018, θα έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης προβλέπουμε ότι και άλλα μέτρα σε σχέση με το χρέος θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μέσω και μάκρο πρόθεσμα εάν χρειαστεί και ε, βεβαίως μετά από επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στα μέσα του 2018. Αναμένει το Eurogroup αυτή η προσέγγιση για τη βιώσιμότητα του χρέους μαζί με την σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στους στόχους του προγράμματος θα βοηθήσει το Δούνου του να κάνει πρόταση έτσι ώστε να συμμετέχει και πάλι πλήρως ε, η δεύτερη αξιολόγηση ε, είναι καθοδόν και ελπίζω στο Eurogroup στις 5 Δεκεμβρίου να έχουμε έκθεση από τις αρχές και τους θεσμούς και ελπίζω και σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων να έχει ε, επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τότε. Μέχρι τώρα έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και αυτό θα επιτρέψει στο Eurogroup να έχει και περαιτέρω συζήτηση για τα μέτρα που χρειάζονται για το χρέος, βράχη πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ε, αυτά και περιμένω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας με χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε Ντάισελμπλουμ, για αυτές τις διαφωτιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις. Θίξατε κάποια βασικά ζητήματα και φαντάζομαι ότι θα εμπαθύνουν τώρα κάποιοι από τους συναδέλφους. Απλώς να σημειώσω ότι προφανώς καταλήξαμε σε διαφορετική φορολογική πολιτική σε επίπεδο CSR και αυτό στο σημερινό μακροοικονομικό πλαίσιο θέτει διάφορα ερωτήματα. Και τέλος πάντων η απόφαση στην οποία καταλήξαμε είναι καλή γιατί δεν είναι νομικά δεσμευτική. Η αναχώραση στάσεως δηλαδή. Η ε, κυρία Ντελάγκη, ευχαριστώ πρόεδρε, θα μιλήσω αγγλικά διότι θα μπορούσα να μιλήσω Ολλανδικά, αλλά ξέρω ότι ο πρόεδρο έτσι κι Αγγλικά θα απαντήσει. Ήθελα να σταθώ στι αναχώρα τάσει και τι πρόσφατε παρατηρήσει τη Επιτροπή, τι ανακοινώσει για τη φορολογική και τη δημοσιονομική επέκταση. Ευχαριστώ για όσα είπατε. Άκουσα πολύ προσεκτικά και τον Ολλανδό Πρωθυπουργό που είπε στο ραδιόφωνο ότι εξέφρασα μια έκκληση για επέκταση σε περισσότερα κρατημέλη, αλλά ε, είπε ότι ήταν κακή η ανάλυση που έγινε κακή ανάλυση από την πλευρά του Επιτρόπου Μοσχοβησί και νομίζω ότι μίλησε και εκ μέρου σα. Το επιβεβαιώνετε. Έτσι είναι. Παρεπιπτόντως, μάλιστα μια νεοφιλελεύθερη πηγή στα ευρωπαϊκά μέσα λέει ότι ίσως και να ε, καλοκοιτάζει τη δουλειά σας ε, ευρωπαϊκά, όχι στα Ε, τέλος πάντων το αφήνω αυτό κατά μέρος. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι εσείς συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση ότι δεν ήταν συνετό να προχωρήσουμε σε δημοσιονομική επέκταση και ότι ο κύριος Μοσκοβισή είπε ότι επειδή το έκανε αυτό, μάλλον ο Επίτροπος Μοσκοβισή είπε ότι θέλει με την κίνηση αυτή να δώσει μια διάσταση Υπουργού Οικονομικών στην Ευρωζώνη ε, με, την, ε, με το συναθρισμένο απολογισμό των στοιχείων. Ξέρω ότι είστε αγωνιστής για τις ε, περαιτέρω κινήσεις στο ΙΔΙΣ και η ερώτησή μου είναι αν πιστεύετε ότι έχουμε ήδη αναλάβει αρκετά βήματα και πόσο μακριά μπορούμε να πάμε, ξέροντας ότι το ΙΔΙΣ και το εθνικό χρέος όπως και εθνική έκθεση ακόμα δεν έχουν επιληθεί ζητήματα. Ευχαριστώ. Ήξερα ότι θα θέσετε την ερώτηση για τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν περίμεναν οι πρώτη σήμερα. Αλλά τι να κάνω, την πάτησα. Η Ευρωζώνη δεν έχει Υπουργό Οικονομικών, έχει 19. Και έχουν μια κοινή συνάντηση και συνεδρίαση που ονομάζεται Eurogroup. Η η Επιτροπή νομίζω ότι έχει δικαίωμα να ε, δίδει συστάσεις σε ένα χώρα και για την Ευρωζώνη συνολικά και για την δημοσιονομική στάση και μετά μπορεί κανείς να συζητά για το κατά πόσον είναι η καταλληλότερη κίνηση. Κάποιοι θα υποστηρίζαν ότι δεδομένες της θέσης στην οποία βρισκόμαστε και στη φάση του οικονομικού κλείσου, κύκλου καθώς τα κενά ε, κλείνουν κάποιες στιγμές, από τις χώρες ίσως να μην είναι συνοτό με τη δημοσιονομική πολιτική να κινητοποιήσουμε περαιτέρω τα πράγματα. Από ε, οικονομική όμω άποψη και στη φάση του οικονομικού κλουμπ που βρισκόμαστε, δεν βρίσκω ότι είναι κακό να έχουμε το Eurogroup. Βεβαίω οι υπουργοί είναι ελεύθεροι να λένε ότι θέλουν. Αλλά αυτό που ανέκαθεν έλεγα στην Επιτροπή και είμαι μεγάλο υποστηρικτή γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι να είναι αυστηρή και σταθερή η Επιτροπή στην εφαρμογή του συμφώνου, εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της, του σεβασμού των κανόνων του συμφώνου και της ε, δημοσιονομικής τάσης, εκεί βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη στάση. Κατάσταση μάλλον. Διότι μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει τάση επέκτασης από δημοσιονομικής σκοπιάς σε χώρες που θα πρέπει αυτή να αξιοποιηθεί, αλλά εκεί θα πρέπει η Επιτροπή να φροντίσει να εφαρμόζονται και τα του συμφώνου. Δηλαδή, με τον καιρό ε, θα πρέπει μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον να πετύχουμε τους στόχους των ε, εξυγιανισμένων ε, προπολισμών. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα. Ούτε μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτή τη δημοσιονομική επιταγή. Αυτό το είδος την κουβέντα λοιπόν θα κάνουμε και στο Eurogroup. Βεβαίως, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός ε, πάντοτε μιλά ε, εκ μου ε, αναγκαστικά εφόσον είμαι Υπουργός Οικονομικών του, αλλά εδώ μιλώ ως Πρόεδρος του Eurogroup. Για το όπως επειδή το αναφέρατε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων, καταθέσεων. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να πιέσουμε για περαιτέρω κάλυψη του κινδύνου. Κάτι που με πρακτικό τρόπο συμβαίνει σε, πολλούς, σε πολλά θεσμικά όργανα ανά την Ευρώπη, όπου τα ζητήματα κάλυψης των περιουσιακών των τραπεζών μπορεί να κάνουν κάποιους να εκνευρίζονται ή να ανησυχούν, αλλά εγώ ησυχάζω όταν βλέπω τέτοιου είδου προβλήματα αντιμετωπίζονται. Και νομίζω ότι το comprehensive package, το σφαιρικό αυτό, το συνολικό πακέτο που έχει προωθήσει η Επιτροπή για την ε, αναχέτηση του κινδύνου είναι γενικώ καλό. Θα το συζητήσουμε και στο Κοφίν και για μερικά ζητήματα. ω Ολλανδός ε, Υπουργός Οικονομικών θα ζητήσω κάπως περισσότερη ισοτιμία. Μεν, αλλά το βασικό είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε προ, να επιτελέσουμε πρόοδο ε, στι προτεραιότητε αντιμετώπισης του κινδύνου. Και σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το ίδιο και δεν κοινή μας δράση. Εδώ χρειάζεται μια ε, κοινή προσέγγιση. Πρέπει να προχωρήσουμε. Και έχω υποστηρίξει ξανά και ξανά ότι για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ε, Οικονομικής Ένωσης και Νομισματικής Ένωσης. Η τραπεζική σταθερότητα είναι επίσης ζωτική σημασία και τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ευρωπαϊκή συνεργασία για το. Πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι θα ολοκληρωθεί αυτό το σύστημα και θα είναι και σταθερό, απαγιωμένο, εδρεωμένο. Χρειάζεται να προβλεφθούν νέε δομέ, νέοι θεσμοί και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Διότι με την επόμενη κρίση που μπορεί να μας πλήξει θα ανακαλύψουμε πόσο είναι δυνατό ή όχι. Πρέπει λοιπόν από τώρα να φροντίσουμε να είναι ισχυρό το οικοδόμημα. Να ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ ενδιαφέρον που παρατηρείτε ότι υπάρχει ανώτατο όριο στα αλλά όχι κατώτατο. Υπάρχει μια έλλειψη συμμετρίας στο σύμφωνο. Υπάρχει το, κατώ, το ανώφλι και δεν υπάρχει το κατόφλι. Τέλος πάντων, μιλάμε εδώ για πλεόνασμα. Πάντως θεωρητικός και όχι μόνο πολιτικός είναι ένα ζήτημα αυτό. Κύριε κυρία Μπερές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέτε ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το όλο σχέδιο που έχουμε ξεκινήσει. Ναι, αλλά σημαντικό είναι να ολοκληρώσουμε και εντός ε, χρονικού διαστήματος εύλογου και αρκετά ε, περιορισμένου, διότι αλλιώς καθυστερούμε. Είπατε ότι μπορεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ του Συμφώνου Σταθερότητα και τη ανάλυση τη δημοσιονομική ε, κατάσταση, τη συναθρισμένη δημοσιονομική κατάσταση τη Ευρωζώνη. Σημαίνει αυτό ότι πιστεύετε ότι κανένα κράτο μέλο δεν διαθέτει απαραίτητη, ε, απαραίτητο περιθώριο για επεκτατική δημοσιονομική πολιτική διότι νομίζω 100% της Επιτροπής δεν μπορεί να, να λάβει δράση σε αυτόν τον τομέα σε όλα τα κατημέλη, μόνο σε αυτούς που έχουν περιθώριο, να αυξήσουν τις δαπάνες τους από τον προπολογισμό. Μια δεύτερη ερώτηση. Αναφέρατε την κατάσταση στην Ελλάδα. Πέραν τη όλη συζήτηση των εμπειρογνωμόνων και τη ανάλυση με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και το κατά πόσο πρέπει να μεθευτεί το πρόγραμμα κτλ. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη ώστε να υπάρξει επιτέλους ανάκαμψη, ανάπτυξη στη χώρα αυτή και επιστροφή των επενδύσεων. Ω προ αυτό δεν θεωρείται ότι ένα σαφές ε, μήνυμα για το θέμα του χρέους, αυτό που περιμένουν τόσο πολλοί επιχειρήσεις για τις επενδύσει και την ανάπτυξη στη χώρα αυτή, είναι κάτι που είναι πραγματικά πολύ αναμενόμενο. Ευχαριστώ. Πρώτα, για το θέμα του περισσότερου περιθωρίου για την αύξηση των δαπανών. Υπάρχουν ένα-δυο κάτι μέλη που σίγουρα έχουν ξεπεράσει τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους και έτσι έχουν περιθώριο να περάσουν λίγο σε περισσότερες δαπάνες. Και είναι λογικό να ε, δαπανίσουν σε εκπαίδευση, σε υποδομέ, στην μελλοντική του αναπτυξιακή ικανότητα. Δεν θα πω ποιε χώρε είναι, αλλά ήδη αυτέ οι χώρε οικονομικά είναι σε καλή θέση. Δεν σημαίνει όμω ότι θα μείνουν και στο μέλλον, εάν δεν ε, προβλέψουν το μέλλον του. Πρέπει να επενδύσουν με ορίζοντα το μέλλον, με προοπτική το μέλλον. Ε, αν δεν μας αρέσει αυτό βέβαια, θα πρέπει να αλλάξουμε το σύμφωνο αλλά το σύμφωνο δεν βάζει όριο για τους μεσοπρόθεσμους ε, στόχους. Οπότε η Επιτροπή έχει εδώ διαφορετικό ρόλο. Είναι μια αρχή με διαφορετική αρμοδιότητα ως προς αυτό. Υπάρχουν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας στο όλο πλαίσιο, αλλά είναι πιο ε, ε, ανοιχτό το θέμα του κατά πόσο χρειάζεται δημοσιονομική επέκταση προς τα έξω νομικά, νομικός μάλλον, είναι πολύ διαφορετική όλη διοργάνωση του θέματος. Το τι είδου επενδύσεις χρειάζονται σε κάθε χώρα. Και σε τι βαθμό είναι άλλο ζήτημα. Πρέπει λοιπόν αυτό να λαμβάνεται υπόψη. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει σίγουρα να το λαμβάνει υπόψη. Και επισήμω η θέση του η αρμοδιότητά τους, η μόχλευση που διαθέτουν ε, για να πιέσουν τα κράτη-μέλη είναι διαφορετική. Είναι πολύ διαφορετικό το αν έχει ξεπεράσει κανείς ή είναι κάτω από τους μεσοπρόθεσμους ε, στόχους. Ασφαλώς. Εγώ δεν αφισβητώ ότι υπάρχει αυτή η ειναι κατω απο τους μεσοπρόθεσμού στοχους ασφαλως εγω δεν αφισβητω οτι υπαρχει αυτη η συσταση Θα το συζητήσουμε στο Eurogroup αν έχει νόημα. Και πώς θα αντιδράσουν σε αυτό οι υπουργοί. Όσοι αισθάνονται ότι τους αφορά το θέμα, έτσι. Είναι μια συζήτηση που θα γίνει στο Eurogroup. Δεν αμφισβητώ το θέμα ότι σωστά το έθεσε η Επιτροπή και το έθεσε επιτάπητος. Έχει ακριβώ το ρόλο να το κάνει αυτό για την Ελλάδα. Το θέμα τη εμπιστοσύνη είναι όντω ζωτική σημασία. Βεβαίω η βιωσιμότητα του χρέου είναι μέρο του κατά πόσο ο παράγοντα εμπιστοσύνη λειτουργεί. Εάν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για την Ελλάδα και του επιχειρηματίε να ε, μπορέσουν να αναλάβουν αυτό το βάρος του χρέους στο μέλλον, το επενδυτικό μέλλον και οι δαπάνες γίνονται πολύ ζωφερές. Πρέπει λοιπόν να μπορεί η Ελλάδα να χειριστεί το χρέος της. Ξέρετε ότι τεράστιος αριθμός μέτρων από το τέλος του 2012 έχουν αναλυθεί. Έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε περισσότερα από το Μάιο στο Eurogroup, πρόθεσμα. Στι 5 Δεκεμβρίου θα υποβληθούν κάποιε νέε προτάσει από την ομάδα εμπειρογνωμόνων και θα γίνουν περισσότερα και προ το τέλο του προγράμματο. Υπάρχει όμω πάντοτε η ερεσιμότητα. Πρέπει να υπάρχει δέσμευση και από τι δύο πλευρέ. Και το λέω στα μέλη του Eurogroup. Χρειάζεται να υπάρχουν υποσχέσει και δέσμευση και από την πλευρά των χωρών πιστοτριών και από την πλευρά τη Ελλάδα για να είμαστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα μπορεί να διαχειριστεί και να αναλάβει τι υποχρεώσει τη. Πρέπει να υπάρχει και η δέσμευση τη ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα αφήσει τίποτα να, τα πράγματα να παρεκτραπούν. Ότι θα συνεχίσει να οικοδομεί ισχυρού θεσμού, μια ισχυρή οικονομία για το καλό τη χώρα, τη Ελλάδα. Και τα δύο σκέλη χρειάζονται για να οικοδομηθεί αυτό το κλίμα εμπιστοσύνη. Uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργη ε, Σταρμπάτη. Κύριε Πρόεδρε, αυτά που μας λέτε τα έχω ακούσει επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο, ότι σιγά σιγά ε, διαφαίνεται η ανάπτυξη, ε, ότι έχει βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση, αλλά ακόμα δεν είναι σταθερή και ότι η Ελλάδα πρόκειται να εφαρμόσει διαρθρωτικές αλλαγές. Χρόνια ολόκληρα τα ακούω αυτά. Το γεγονός όμως είναι ότι η Ευρωζώνη είναι η ζώνη εκείνη η οποία αναπτύσσεται λιγότερο από πουδήποτε και οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Και ε, το λόγο το ξέρουμε. Δεν είναι ότι το ευρώ είναι υποτιμημένο. Η δική μας Επιτροπή Προπολογισμών έχει ε, παρουσιάσει μια, ένα, ε, ένα πλάσιο πολυψισμό, έχουμε μια ισοτιμία που για μας ε, είναι σταθερή και αυτό που κάνουμε είναι αυτό που λέει ο Κένς ε, bigger my neighbor policy όμως αυτά τα οποία γίνονται τώρα αυτά ήταν η θελημένα μέσα στην Ευρωζώνη και τώρα ξαφνικά ακούω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αν η Γερμανία είναι λιγότερο ανταγωνιστική, δηλαδή αν η Γερμανία κάνει τα ίδια λάθη που έκαναν άλλες χώρες και τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κοιτάξτε, στην ε, Ευρωζώνη λένε πολύ πρέπει να υπάρχει ισορροπία και λένε ότι αυτά πρέπει να κάνει η Γερμανία. Εσείς πιστεύετε ότι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ του να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα της Γερμανίας και με τον τρόπο αυτό να πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουμε τα προβλήματα της Ευρώπης. Πιστεύετε ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρωζώνη με το να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα της Γερμανίας. Απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερωτήσή σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω το εξής. Υπάρχει μια τάση, όχι μόνο στην Ευρώπη, θα έλεγα γενικότερα για μια ρεαλιστική πολιτική. Πρέπει δηλαδή κανείς να γνωρίζει τα γεγονότα, τα γνωρίζει και μετά λέει το αντίθετο. Και η αλήθεια είναι ότι για τέταρτη κατά σειρά ετός βελτιώνεται η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και επίσης μια σειρά χωρών έχουν να επιδείξουν μεγάλη ανάπτυξη. Εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν αρκετές διαφορές και εξακολουθεί να ισχύει ότι μεσοσταθμικά η ανάπτυξη ανέρχεται σε 1,6% ίσως φέτος να είναι κατά τη μεγαλύτερη. Είναι επίσης γεγονός ότι τα ελλείμματα θα μειωθούν στο κάτω από 2% μεσοσταθμικά πάλι στην Ευρωζωνική. αυτά είναι στοιχεία. Δεν σας τα λέω γιατί θέλω οτιδήποτε να εξοραίσω. Είναι στοιχεία. Επί τη βάση λοιπόν αυτών των στοιχείων ας δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι αλήθεια ότι έχουμε τη μικρότερη ανάπτυξη στον κόσμο όπως είπατε εσείς. Μα δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Και δεν ξέρω γιατί το είπατε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το είπατε τα στατιστικά δεδομένα το λένε αυτό, λέει ο Ευρωβουλευτή. Ναι, αλλά δεν είναι αλήθεια. Ξέρω ότι θα, λέει ο κύριο Ντάζελμπλουμ, ξέρω ότι το είπατε αυτό γιατί μετά θέλετε να πείτε ότι για όλα αυτά φταίει το ευρώ. Αλλά όπως είπε και ο Στίγκλιτς, ε, για όλα τα προβλήματα μπορεί κανείς να κατηγορεί το ευρώ. Αυτό όμως δεν είναι η σωστή ανάλυση. Η ανάλυση είναι ότι υπάρχουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας σε πολλές χώρες, ότι χτυπηθήκαμε από κρίση, πάρα πολλοί δημοσιονομικοί τομείς, προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτό, δηλαδή η αναμόρφωση και ανασύσταση των τραπεζών συνεχίζεται όλα αυτά τα γεγονότα και οι κινήσεις θεωρώ ότι βαδίζουν προς τη σωστή κατάπτυνση. Εάν τώρα εσείς θέλετε να ρίξετε το βάρος στο ευρώ, μπορείτε να το κάνετε. Ε, δεν νομίζω όμως ότι η σταθερότητα πριν από το ευρώ ήταν τέλεια, αλλά από ό,τι φαίνεται έχετε κοντή μνήμη. Δεν θυμάστε καλά. Τώρα, λέτε ερώτηση, ρητορική, η Γερμανία να έχει χειρότερη ανταγωνιστικότητα. Όχι, φυσικά, εμείς δεν λέμε τέτοιο. Δεν λέμε ότι ε, θα μπορούσαν να επιτύχουν τα προγράμματα ανάκαμψης μόνο αν η Γερμανία χάσει την ανταγωνιστικότητά της. Η Γερμανία σε μεγάλο βαθμό εξάγει εκτός Ευρωζώνης. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Και εγώ πιστεύω ότι από κοινού μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και είναι πολύ δύσκολη γιατί χτυπηθήκαμε από βαριά κρίση ε, αλλά συνεχίζεται η διαδικασία. Ας είμαστε πιο κοντά σε γεγονότα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία αισιοδοξίε και ε, υπάρχει και κάποια αποφασιστικότητα να επιμείνουμε στην ανάπτυξη. Παρεπιπτόντος, ε, η Γερμανία πάνω από το 3% είναι αρκετά χρόνια, αλλά αυτό δεν μοιάζει να επηρέασε την ανταγωνιστικότητά τους και να περάσουν οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Κόρα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, Γερόν. Θα ρωτήσω αγγλικά, όχι ολλανδικά, γιατί έτσι κι αλλιώς αγγλικά θα απαντήσεις, το ξέρω. Θέλω να ρωτήσω και κάτι για τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το μισό δισεκατό ε, του ΑΕΠ, δηλαδή 50 δις ευρώ, θα πρέπει να επενδύονται από χώρες που έχουν το περιθώριο αυτό. Και εξ όσων γνωρίζω αυτές οι τρεις χώρες είναι Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γερμανία. Ε, η Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία που τη γνωρίζεις πολύ καλά υπολόγισε ότι αν οι χώρες αυτές αξιοποιήσουν όλο το περιθώριο που έχουν ε, στις συστάσεις ε, θα επενδύσουν 0,29%. Καμία σχέση με τα 50 δις ε, για τα οποία μιλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι βγάζεις από αυτό το συμπέρασμα. Ε, συμφωνείς ότι υπερβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας ότι θα πρέπει να επενδυθούν 50 δις επιπλέον. Και δεύτερη ερώτηση. Μια δήλωση έκανε πρόσφατα ο Σόιμπλε, Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, και είπε ότι θα πρέπει να είναι ε, πιο ανεξάρτητη η αρχή αυτή που θα επιβάλλει τα δημοσιονομικά και δεν θα υπόκειται σε διάφορα συμφέροντα. Θα με ενδιαφέρε, θα ήταν καλύτερη ε, μια ανεξάρτητη αρχή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει αυτό τον ρόλο. Για το πρώτο θέμα, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερβάλλει στις συστάσεις, Αναφέρθηκα και προηγουμένως αυτό. Η σύσταση για μια δημοσιονομική επέκταση ε, και ε, η τήρηση του συμφώνου ε, είναι πράγματα κάπως αντιφατικά μεταξύ τους. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο σωστά. Η πρώτη ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διατηρηθεί το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη που κρατάει ενωμένη την Ευρωζώνη. Δεν το λέω αυτό επειδή είμαι κανένα σκληρό καλβινιστή από την Ολλανδία. Κατά τα άλλα, ξέρετε ότι είμαι και καθολικό. Αλλά ε, τα ζητώ διότι ξέρω από την εμπειρία μου στο παρελθόν πόσο σημαντικό είναι να διαφυλάσσεται η ε, αξιοπιστία του συμφώνου. Και υπάρχει ένας πειρασμός να χαλαρώνει κανείς σε καλούς καιρούς και μετά όταν έρχονται οι ε, χαλεποί καιροί να τα λαμβάνουμε πιο σοβαρά υπόψη. Αυτή είναι η εμπειρία του παρελθόντος. Ας βεβαιωθούμε ότι θα ε, διατηρήσουμε ενωμένη την Ευρωζώνη σε σταθερή κατάσταση. Ε, δεύτερον, για την ανεξάρτητη υπηρεσία θυμίζω την έκθεση των πέντε προέδρων όπου έλεγαν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο ας πούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να εκτιμά και να αξιολογεί που βρίσκονται οι κυβερνήσεις και οι εθνικοί προϋπολογισμοί σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους στο σύμφωνο. Δηλαδή αυτοί να δίνουν τα στοιχεία και τα δεδομένα και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία να παίζει το ρόλο που της αναλογεί για την ε, εκτέλεση και την εφαρμογή και η ε, επιβολή ακόμα εάν τα κράτη-μέλη δεν συμμορφώνονται προς τους κανόνες αυτούς. Αυτό πρότειναν οι πέντε πρόεδροι στην έκθεσή τους και εγώ παραμένω υπέρμαχος αυτής της πρότασης. Έχει συσταθεί αυτό το Συμβούλιο υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, τώρα γίνεται μια συζήτηση είναι αρκετά ανεξάρτητο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το Δεκέμβριο θα έρθει για πρώτη φορά ο Πρόεδρος. Ελπίζω να προσεκλήθη, δική μου ε, πρόθεση για να δούμε πώς βλέπει το δικό τους ρόλο και πώς μπορεί να προχωρήσει η συνεργασία μας. Ρομπέρτο, Ρομπέρτ, έχω και άλλη ερώτηση συμπροματική λέει κόρα. Την περασμένη εβδομάδα είχε έρθει ο κύριος Γεωργίου της Ελστάτ ε, στην ομάδα εργασίας μας και μας είπε ότι πήγανε κάποια πράγματα στραβά στην Ελστάτ με τις στατιστικές. Τώρα οι στατιστικές που παίρνετε από την Ελλάδα είναι απολύτως αξιόπιστες. Ε, ο, ο, ο επικεφαλής της Eurostat αυτό μας έχει δηλώσει. Απάντησε. Πολύ ε, προσοχή χρειάζεται όταν ρωτάτε ένα πολιτικό αν μπορεί να εμπιστεύεται τις στατιστικές. Γιατί ό,τι και να πω θα μπορούσε να βλάψει την ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών μας δεν αναπόκειται σε μένα να το αξιολογήσω. Η Eurostat το κάνει αυτό. Κατά πόσο οι εθνικές στατιστικές αρχές κάνουν την σωστή δουλειά και με την ποιότητα που θέλουμε εμείς. Έτσι κι αλλιώς ό,τι και να σας πω, δεν θα με πιστέψετε να σας πω ότι ε, οι εθνικές στατιστικές της Ολλανδίας είναι καλές ή κακές. Θα μου απαντούσατε εσύ πολιτικός είσαι, δεν είναι δική σου δουλειά. Αυτό λέω ακριβώς. Μην ε, ε, καθιστάτε υπεύθυνου για τις στατιστικές του πολιτικού. Θα πρέπει να έχουμε ε, υψηλού επίπεδου στατιστικές σε όλη την Ευρώπη και μετά ε, με βάση αυτές να κάνουμε πολιτική συζήτηση και να διαφωνήσουμε. Αλλά τα στοιχεία είναι στοιχεία και θα πρέπει να τα ε, γνωρίζουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Παπαδημούλης, παρακαλώ. Thank you, Chair. Mr. Dasselum, Κύριε Ντάσερμπλουμ, θα μιλήσω ελληνικά, παρακαλώ. Θα ήθελα πριν απ' όλα να ενημερώσω τη συνάδελφο που ρώτησε προηγουμένως ότι πριν μια ακριβώς βδομάδα, και το λέω και στον κύριο Ντάισεμπλουμ, ήταν εδώ ο κύριος Ραντερμάχερ, ο επικεφαλής της Eurostat, Γερμανός. Τον ρωτήσαμε για την ποιότητα των δημόσιων στατιστικών σήμερα στην Ελλάδα. Μας είπε ότι έχει σημειωθεί σημαντικότατη πρόοδος, ότι τα μαγειρέματα αφορούν μια περίοδο του παρελθόντος, ότι δεν συμβαίνουν τώρα και ότι τώρα το μόνο που θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει είναι διοικητικέ αδυναμίες, όπως υπάρχουν σε όλες τις εθνικές στατιστικές, αλλά όχι πολιτικές παρεμβάσεις. Και νομίζω ότι δεν πρέπει αυτή την ώρα που χρειάζεται εμπιστοσύνη να παίζουμε με αυτά τα θέματα. Κύριε Ντάισελμπλουμ, σας καλωσορίζω και σημείωσα με προσοχή τις θετικές σας δηλώσεις για την Ελλάδα. Αναφερθήκατε σε σημαντική πρόοδο από το Φεβρουάριο, σε εντυπωσιακό κατάλογο μέτρων που έχουν ληφθεί, στην ανάγκη να οικοδομηθεί ακόμη περισσότερο εμπιστοσύνη και δηλώσατε και αισιόδοξο ότι μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου ελπίζετε να υπάρχει το περίφημο staff level agreement σε επίπεδο υπηρεσιακό. Θα έχετε υπόψη σας και το μύθο του Σισίφου. Οι Έλληνες τηρούν τις δεσμεύσεις τους και περιμένουν και από τους δανειστές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Χθες ο κύριος Δράγκη, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, μίλησε για την ανάγκη αυτό το θετικό momentum να μην χαθεί, αλλά να αξιοποιηθεί και να μην έχουμε αναβολές και καθυστερήσεις. Σας ερωτώ λοιπόν, τι μπορούμε να περιμένουμε από το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου όσον αφορά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης σε συνδυασμό με τα μέτρα ελάφρυσης του χρέους και με τα, πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018. Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των δανειστών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά δραστικότερα μέτρα ελάφρυσης του χρέους και αποσαφήνισή τους από τώρα και για τα μεσοπρόθεσμα και επίσης ζητάει χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα για την Ελλάδα μετά το 18 προκειμένου να έχουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη. Η ερώτησή μου είναι τι βήματα είσαστε διατεθειμένοι να κάνετε ως Eurogroup προκειμένου να πετύχετε μια συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτά τα δύο θέματα. Σας ευχαριστώ. Thank you. Um... Ευχαριστώ τι μπορούμε να αναμένουμε στις 5 Δεκεμβρίου στο Eurogroup. Θα ακούσουμε τους θεσμούς και ελπίζουμε να υπάρχει συμφωνία staff level agreement για τη δεύτερη εξολόγηση Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να ε, έχουμε μια ισχυρή βάση για να προχωρήσουμε. Για να γίνει μια καλή συζήτηση. Δεύτερο θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια από τα στοιχεία που παραμένουν σε εκκρεμότητα από προηγούμενες συμφωνίες το ένα είχε να κάνει ε, με το πλεόνασμα, το πρωτογενές, 3,5 ε, είναι αυτό για το 2018 και είμαστε σε αυτό το δρόμο και σε προηγούμενη συμφωνία αναφέρεται το μέσο πρόθεσμο. Πόσο μακριά είναι το μέσο πρόθεσμο ε, ως στόχος. Αυτό θα συζητηθεί. Ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι δεν μπορείτε να ζητάτε από την Ελλάδα να το διατηρήσει αυτό για πολύ μεγάλο διάστημα. Άλλοι λέγουν ότι θα είναι απαραίτητο δεδομένο ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συμμορφωθεί με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Άρα ε, και αυτό προβλέπει αρκετά σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα. Και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ότι ε, η Ελλάδα ε, απομακρύνεται και εγκαταλείπει το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να βρούμε ένα ρεαλιστικό δρόμο να προχωρήσουμε. Και λέω ρεαλιστικό γιατί πιστεύω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει και κάποιο δίκιο. Όταν σου λέει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% για τεράστιο χρονικό διάστημα είναι ε, ε τεράστιο στόχος και υπερβολικό να το ζητάμε και θα πρέπει να παραμένουμε ρεαλιστές σε αυτό το επίπεδο και αυτό θα ε, έχει να κάνει και με την ε, βιωσιμότητα του χρέους για ε, μακρύ χρονικό διάστημα. Όπως σας είπα, θα ακούσουμε τι θα μας πει στις 5 Δεκεμβρίου ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο ESM, τι μπορούν να κάνουν βράχη πρόθεσμα για να μειωθεί το κόστος διαφόρων δανείων κτλ. Τι μπορεί να κάνει ο ESM, εκεί είμαι αρκετά αισιόδοξο. Έχουμε απελευθερώσει για το 2018, μέχρι το 2018 ε, επιπλέον μέτρα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, θα ρωτήσει πόσο προσιλωμένοι είστε εσείς σε αυτή την προσπάθεια. Ε, είναι εύλογο το ερώτημα, θα το συζητήσουμε αυτό και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει συμφωνήσει ήδη το Μάιο, όπως είπαμε, πριν τα τέλη του έτους να πάει στο Διοικητικό του Συμβούλιο όπως είπε και ο Μάριο Ντράγκη, να βασιστούμε σε αυτή τη θετική ατμόσφαιρα και την επικοδομητική που επικρατεί αυτό τον καιρό, να μην την αφήσουμε να μας ξεφύγει, να κάνουμε βήματα πρόοδου, βήμα-βήμα θα γίνει αυτή η προσπάθεια. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι το δικό μου στυλ, βήμα-βήμα. Ορισμένοι θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα, άλλοι μπορεί να τα έχουν στυλώσει τελείω. Ε, θα προχωρήσουμε, αλλά βήμα-βήμα. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Δεν πρέπει να κατηγορείτε το ευρώ το ίδιο για την αργή ανάπτυξη, αλλά η έλλειψη συνεκτικής και συνεπούς ε, χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με το κοινωνόμισμα. Και μετά βλέπουμε το παραμύθι σας των μεγάλων αυτών επιτυχημένων μέτρων, θα πρέπει να κρυθεί και με πρίσμα την στάση της ε, ΕΚΤ και των χαμηλών επιτοκίων που διαρκώς ε, πιέζουν τις ασφαλίσεις μας, τα συνταξιδοτικά μας και το Ολλανδικό συνταξιδοτικό, έτσι, και την πραγματική οικονομία και τις τράπεζες που λειτουργούν εντός αυτής. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη κοινή ε, δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής. Και επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώς έλαβε ένα θετικό βήμα με το κοινό δημοσιονομικό περιθώριο. Εσείς θα το στηρίξετε αυτό. Δεν ήταν σαφές στις εσωτερικές σας παρατηρήσεις. Και δεύτερον, η Ολλανδική κυβέρνηση μπορεί να κάνει κάτι για να βελτιώσει τη συνοχή τη συνεκτικότητα της κοινή οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης και να σταματήσει να παρεμποδίζει τα μέτρα ή την καταπολέμηση του φορολογικού ανταγωνισμού στην Ευρώπη στις 18 Νοεμβρίου αποστήλατε επιστολή προς το Ελλανδικό Κοινοβούλιο για να ζητήσετε πενταετή αναβολή τη οδηγία για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Και ε, επισήμω η Ολλανδική κυβέρνηση έχει ταχθεί κατά το ΕΚΤ και ζητά να χαμηλώσουν τα επιτόκια για τι επιχειρήσει. Και εσεί αργείτε για να εφαρμόσετε και τι αποφάσει του, του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία. Από τι 13 Ιουνίου έπρεπε να υλοποιηθούν και ακόμα λέτε ότι θα γίνει του χρόνου. Ποιο είναι ο λόγο ε, των προγειοοικονομικών ε, τη Ολλανδία, λοιπόν. Αυτά θα ήθελα να ξέρω. Το καλό είναι ότι είμαι μόνο ένας. Και πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο. Η άποψή μου για την ε, σύσταση, για την ε, δημοσιονομική αποτίμηση της Ευρωζώνης. Νομίζω ότι είναι γεγονός. Κάποιες χώρες έχουν δημοσιονομικό περιθώριο και θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για να επενδύσουν συνετός. Όμως, οι εθνικές κυβερνήσεις θα αποφασίσουν σε τι βαθμό θέλουν να επενδυθούν αυτά τα ποσά και πώς. Νομίζω με τον καιρό, αν και τα πράγματα πάνε αρκετά γρήγορα, και άλλες χώρες θα, βρεθούν, θα σε αυτή τη θέση. Σε θέση όπου θα μπορούν να κοιτάξουν το μέλλον με αισιοδοξία περισσότερο και να συζητήσουν τις μελλοντικέ τους επενδύσεις αντί απλώς να κοιτάζουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κρίση. Αλλά αυτό θα αποφασίσουν τα κάτι μέλη. Δεύτερον, για τα φορολογικά με συγχωρείτε που λυπάμαι που έχετε τόσο απογοητευτεί, αλλά ως πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ πρέπει να πω ότι πολύ μεγάλη πίεση ασκήσαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βρεθεί λύση για τα φορολογικά. Είτε σας αρέσετε όχι, νομίζω ότι αυτά που έχουν γίνει ως τώρα είναι μεγάλο βήμα και η Ευρώπη ήδη είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή της συμφωνίας BEPS. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε το Δεκέμβριο και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία τον ε, Δεκέμβριο στο ΕΚΟΦΗΝ. Τώρα, αν η Ολλανδική κυβέρνηση έχει συγκεκριμένε επιθυμίε για το θέμα αυτό, ναι, όλοι έχουμε. Ναι, αλλά θέλετε να εφαρμοστεί πέντε χρόνια καθυστερημένα όπω κάψετε στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο ή όχι. Γιατί αυτά που μα λέτε δεν συνάδουν απολύτω με αυτά που λέτε στου Ολλανδού ε, συναδέλφου στο Βουλή. Θέλετε να αναβληθεί για πέντε χρόνια. Θέλω συμφωνία το Δεκέμβριο η εφαρμογή αυτού του σκέλους για τις ε, υβριδικές ε, ε, λήψεις αντιστοιχήσεις με τρίτες χώρες θα χρειαστεί χρόνο. Θα χρειαστεί εξυγίανση και αναδιάρθρωση κάποιων εταιριών. Ω Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών θα ζητήσω περαιτέρω χρόνο, όπω και άλλε χώρε ζήτησαν περαιτέρω χρόνο για μετάβαση σε κάποια άλλα ζητήματα. Για τι χρειάζονται χρόνο για να γύρει σωστά η εφαρμογή και να επιτελεστεί πρόοδο. Ναι, αλλά πενταετή αναβολή σημαίνει βασικά ότι συνεχίζεται να υποφελείστε τα κέρδη των ε, πολυεθνικών. Πέντε χρόνια αναδιάρθρωση λέτε. Αυτό χρειάζεται. Και μήπω κοιτάζετε το συμφέρον σα ω Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Κανένα πρόβλημα. Διαρκώ είμαι και Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών. Γιατί στι κάτω χώρε αυτό απασχολεί και συζητιέται. Δεν είναι κατά του προσώπου σα, είναι επί τη ουσία. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ω Υπουργό Ω Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών, θα υποστηρίξω ότι το σημαντικό είναι να υπάρξει συμφωνία το Δεκέμβριο και να ε, επιτελεστεί πρόοδο σε όλα αυτά τα φορολογικά ζητήματα. Έχω δεσμευτεί την τελευταία διετία να επιτελεστεί εδώ πρόοδο και μπορείτε να με επικρίνετε που δεν έχω κάνει αρκετά Ξέρω ότι στην Ολλανδία το θέμα αυτό είναι καυτό, αλλά θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και να επιτελούμε πρόοδο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπέατριξ από την EFTD με κύριε Ντάσιλμπλουμ, ε, τα δημόσια οικονομικά της ε, Ευρωζώνης ε, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Νομίζω ότι συμφωνούμε από αυτού και το έλλειμμα στην Ευρωζώνη από 1,8 εφέτος πρέπει του χρόνου να κατέβει στο 1,5%. Αυτό ακούγεται πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Όσον αφορά την ανάπτυξη, το χρέος, τα ελλείμματα, αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το σύμφωνο σταθερότητας είναι αν θέλετε ένας γενικό κανόνας έτσι ώστε να παραμένει σταθερό το χρέος ενός κράτους από 16% αν έχει ένα κράτος χρέος 16% ε, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχει την ίδια περίοδο η ανάλογη ανάπτυξη έτσι ώστε το χρέος να είναι βιώσιμο. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία. Με, αλλιώς να το πούμε, εάν το χρέος αυξηθεί κατά 5% τότε το ΑΕΠ θα πρέπει και αυτό να αυξηθεί κατά 5% κατά το ίδιο ποσοστό. Φτάνουμε λοιπόν στα πραγματικά προβλήματα της Ευρωζώνης. Το 2016 το χρέος ανέρχεται σε 91,6% του ΑΕΠ που αυτό σημαίνει έλλειμμα και επίση έλλειμμα 1,8%. Θα αυξηθεί περαιτέρω το χρέο κατά 2%. Εξ αυτών ε, προκύπτει το αίτημα προ την ανάπτυξη, θα πρέπει να είναι εξίσου μεγάλη, όμω η πιθανή ανάπτυξη τη Ευρωζώνη προβλέπεται ότι θα ανέλθει μόνο σε 1%. Και διαβάζω στην ισοσελίδα τη ε, ΕΚΤ του Απριλίου του 2015 ε, αναφέρει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΠ ότι το ενδεχόμενο μάλλον Αλλιώς, οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν ποσοστό ανάπτυξης που θα είναι κάτω από 1% ε, το χρόνο στην Ευρωζώνη. Άρα δηλαδή το δυναμικό ανάπτυξης είναι κάτω του 1%. Με άλλα λόγια, η Ευρωζώνη ήδη βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση και βραχυπρόθεσμα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εξωτερικοί παράγοντες όπως το πρόβλημα των Ιταλικών τραπεζών, το δημοψήφισμα στην Ιταλία. Αυτά είναι εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά. Και ρωτώ, μήπως θα θέλετε να έχετε καλύτερη άλλη δουλειά να κάνετε άλλο επάγγελμα ενώ από αυτό που έχετε τη στιγμή. Δεν θα προτιμούσατε να ασκείτε άλλο επάγγελμα από αυτό που ασκείτε τώρα. Κύριος Ντάισελμπλουμ, κοιτάξτε, ε, Πρέπει καταρχήν να κατανοήσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το δυναμικό ανάπτυξη στην Ευρωζώνη δεν θα ξεπεράσει ποτέ το 1%. Αλλά ήδη υπάρχει μεσοσταθμικά ανάπτυξη 1,6% και αυξάνεται συνεχώς. Ε, μία μεγάλη χώρα κρατών είναι γύρω στο 2% και κάποιες άλλες είναι γύρω στο 1%. Όμω περίπου όλε οι χώρε ξεπερνούν αυτό το δυναμικό ανάπτυξη, ε, όπω το αναφέρατε εσείς.

Άρα δηλαδή τι σημαίνουν όλα αυτά. Τα ελλείμματα μειώνονται όλο και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Όλο και περισσότερε χώρε τα επόμενα δύο χρόνια θα επιτύχουν του στόχου, του μεσοπρόθεσμου, του ε, δημοσιονομικού και έτσι και όλο και περισσότερε χώρε ε, θα επενδύσουν. Μέχρι τώρα πράγματι ε, οι χώρε, αρκετέ χώρε χτυπήθηκαν από την κρίση και αυτό ο αρνητικό κύκλο θα αντιστραφεί σε θετικό. Τα χρέη θα μειώνονται σε όλο και περισσότερε χώρε. Αυτό βέβαια χρειάζεται χρόνο. Αν υπάρχει κρίση προϋπολογισμών ε, χρειάζεται χρόνος για να ρυθμίσει κανείς το χρέος. Δεν υπάρχει μαϊκή συνταγή. Αν την έχετε πέστε τι μου. Δεν υπάρχει μαϊκή γρήγορη συνταγή για το δημόσιο χρέος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να τακτοποιήσουμε τα ε, δημόσια οικονομικά μας ε, διότι πράγματι πρέπει να δούμε να μην αυξηθούν τα δημόσια χρέη ε, κατά το μέλλον στον ίδιο βαθμό. Στους προϋπολογισμούς μας πλέον υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες απορρόφησης κραδασμών. Όμως δεν υπάρχει ταχεία ρύθμιση του χρέους. Ε, δεν μπορούμε και τους προϋπολογισμούς και την ανάπτυξη να τα ρυθμίζουμε κατά μια χρονική περίοδο και το χρέος και ονομαστικά και ως ποσοστό του ΑΕΠ να αρχίσει να μειώνεται. Αλλά τέλος πάντων κάπως βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας έλεγα να διαβάσετε το 162, το Β, αυτό το άρθρο, για να δείτε τι ακριβώς αναφέρεται εκεί σχετικά με το έλλειμμα που τα ανέφερε ε, και ο κύριος Ντάσελμπλουνκ, ο Γκέρολ Άνεμανς. Από την ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ντάσελμπλουνκ, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ρωτάτε, σε δύο, και μάλλον τι εννοείτε, σε δύο περίεργες ε, συνεντεύξεις που δώσατε την περασμένη εβδομάδα. Το ένα ήταν για την εφημερίδα Τράου, πίστη και το άλλο σε ένα κανάλι RTL ε, τηλεόραση. εκεί παραδέχεστε ότι η Ολλανδική κυβέρνηση στην πιο βαθιά ε, κρίση του ευρώ, πώς το είπατε, ε, και εξέτασε και το ενδεχόμενο να ε, μην επιβιώσει το ευρώ. Εδώ που είμαστε μια ανοιχτή δημοκρατία θέλω να σας ρωτήσω τι μοντέλο σκέφτεστε. Ε, θα επανέλθετε στο ε, παλιό νόμισμα δηλαδή το φλωρίν και ποια είναι τα έγγραφα που έχουν κυκλοφορήσει ε, για να προετοιμάσετε την περίοδο μετά το ευρώ. Αυτό ήταν για το RTL και στην εφημερίδα Τραού πίστη ε, ορίζεται την ποιότητα του ευρώ. Ε, είναι ένα νόμισμα που μοιάζει περισσότερο με το παλιό Ολλανδικό ή με το γερμανικό Μάρκο ε, και λιγότερο με την Ιταλική Λιρέτα. Τι συγκρίσεις είναι αυτές γεωγραφικές, περιφερειακές για μένα. Ε, μπορεί να φαίνεται λογικό, αλλά για εσά που είστε πρόεδρος της Ευρωζώνης και του Eurogroup, είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα. Ε, δηλαδή, αν είναι ένα κοινωνικό μοντέλο κορσές που πρέπει να εφαρμόζεται παντού για να είναι σταθερό το ευρώ, ε, λέτε ότι αυτό θα πρέπει να είναι ολλανδικό-γερμανικό μοντέλο. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να μιλάτε με τέτοιο τρόπο. Δεν καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ που διαβάζετε όλες μου τις συνεντεύξεις και τις βλέπετε. Ναι. Ε, δουλειά μου είναι. Δουλειά σου είναι. Με χαρά θα ήθελα να κάνω κι εγώ αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, πρώτη παράθεση, δεν την αναγνωρίζω, δεν τα είπα έτσι στην RTL, για τη δυνατότητα να μην επιβιώσει το ευρώ. Πρώτον, δεν ήμουν υπουργό τότε που συζητήθηκε αυτό, για ποιο ήταν το εναλλακτικό μοντέλο. Είναι γεγονός ότι το υπουργός, ε, ο υπουργό και η τότε κυβέρνηση ε, είναι ερώτηση ε, προετοιμαζόσαστε γι' αυτό, ήμασταν στη χειρότερη κρίση και η Ολλανδική κυβέρνηση ε, ε, το εξέτασε και αυτό το ενδεχόμενο. Θέλουμε να διατηρήσουμε το ενιαίο νόμισμα, αλλά εάν δεν πετύχει, τι θα γίνει. Ντάισελμπρουμ λέει εδώ, εσείς απαντήσατε. Δεν ξέρω. Αυτά λέει η RTL. On quote και στην τηλεόραση μπορείτε να το δείτε. Ε, να χαίρομαι που παραθέσατε το σύνολο, γιατί αυτό έδειξε πόσο ε, Προσιλωμένο είμαι στη διατήρηση ε, της Ευρωζώνης, στην ακαιρεότητα και στην ενότητά της και να ενισχύσουμε αυτό που έχουμε και να ε, οικοδομήσουμε από αυτού παρά να συζητούμε ή να ξανανοίγουμε πράγματα που μπορεί να είχαν συζητηθεί στο παρελθόν. Τώρα, όταν ήμασταν πραγματικά στην πιο βαθιά κρίση Ευρωζώνης, του ευρώ, πολλέ κυβερνήσει αναρωτήθηκαν τώρα τι θα απογίνει και τι θα κάνουμε. Αλλά ποτέ δεν κυριάρχησε αυτό η συζήτηση, ούτε ήταν ε, στο προσκήνιο τη παρούσα ή τη προηγούμενη ή άλλων Ολλανδικών κυβερνήσεων. Κατά τα άλλα, είναι πολύ παλιά αυτή η ε, συνέντευξη. Ε, πόσες παλιές ακόμα παλιε ακομα συνεντεύξει μου θα μου βγάλετε. δεύτερον, για το ευρώ. όταν μίλησα για το ευρώ, συγκεκριμένα αναφέρθηκα στο πόσο αξιόλογο είναι να έχεις ένα ισχυρό νόμισμα το οποίο να εμπιστεύονται και σταθερό. Και υπό την έννοια αυτή το συνέκρινα με κάποια παλιά νομίσματα. Δεν ε, θέλουμε να έχουμε ένα γερμανικό ή ολλανδικό μοντέλο για την Ευρωζώνη ή κανένα άλλο μοντέλο. Έχουμε ορίσει ένα κοινό πρότυπο που ακολουθούμε και τμήμα αυτού βασίζεται στην δημοσιονομική σταθερότητα και την ισχύ και επίσης αντιμετωπίζουμε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μακροοικονομικές ισορροπίες. Άλλο και είναι, είναι να έχουμε μια κοινή νομισματική πολιτική. Αυτό το μοντέλο επιλέξαμε και όχι κάποιο συγκεκριμένο. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριος Νίδερμαγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα, πρόγραμμα, σε ένα στοιχείο του προγράμματός σας, μια διεθνή διάσταση που συζητάει το Eurogroup. Πρώτον, ποιοι είναι οι εξωτερικοί κίνδυνοι ε, κατά την άποψή σας για την Ευρωζώνη και την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και δεύτερον, σε ποιο βαθμό, πώς να το πω, μια πιο σκληρή τάση των Ηνωμένων Πολιτειών στα εμπορικά ζητήματα και την Κίνα μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Και τέλος, πώς βλέπετε την πρόοδο στην Κίνα, στη μείωση των ε, υπερβολικών πλεονασμάτων έχουν και των κρατικών ενισχύσεων και την ενδεχόμενη χειραγώγηση του νομίσματος. Ε, και ένα τελευταίο για τα φορολογικά. Παρά το γεγονός ότι απογοητεύτηκα λίγο από τις απόψεις που έχετε για το πώς θα επιτευχθεί πρόοδος, γιατί αν έχει ορίζοντα πενταετίας, ε, νομίζω ότι δεν ε, επιτυχάνεται καμία πρόοδος. Σε ποιο βαθμό το έχει συζητήσει αυτό το Eurogroup για το πακέτο για το κοινό αναποιημένο ε, σύστημα φορολογικής βάσης. πρόεδρε, για να καταλάβω καλά και να διαλύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Το Eurogroup δεν συζητάει, πόσο μάλλον δεν αποφασίζει τα φορολογικά καθόλου. Καθόλου δεν το συζητάμε. Αυτά που μας είπατε θα συζητάει το ECOFIN το Δεκέμβριο και τους επόμενους μήνες, όχι το Eurogroup, ε, για τους εξωτερικούς κινδύνους. Παραμένουν πολλοί. Αλλά θα ήμουν πιο αισιόδοξο αυτή τη στιγμή για την Κίνα από ε, σε σχέση πριν από ένα-δύο έτη. Βεβαίω έχουν πλεονάσματα σε πολλού τομεις τη οικονομία, αλλά προχωρούν στι μεταρρυθμίσει και εκείνοι. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν και πιστεύω ότι έχει δίκιο η Ευρώπη να απαντά σε αυτά και να προστατεύει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ε, σε αυτού του κλάδου τη οικονομία. Πάντω, οικονομικά, ε, εγώ θα ήμουν πιο αισιόδοξο. Κάνουν εκεί μια μεταρρύθμιση, ένα μετασχηματισμό που πηγαίνει αρκετά καλά. Η Αμερικανική κυβέρνηση και βέβαια ε, παραμένει το μέγα ερωτηματικό για μας. Νομίζω είναι δίκαιο να προξοφλήσουμε ότι θα αποτελματωθούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις, χωρίς να μας χαροποιεί αυτό. Πάντως αυτό μπορεί να αποδειχθεί χαμένη ευκαιρία. Το συντομότερο θα το θέσουμε. Αυτά είναι τα βασικότερα ζητήματα που ρωτήσατε, νομίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Στάνη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να θίξω ένα από τα ζητήματα για τα οποία θα χρειαστεί περισσότερη σαφήνεια στο τέλος του μήνα. Η δουλειά της Επιτροπής της Βασιλείας ένα από τα ζητήματα επιτάπητος είναι η χρήση των εσωτερικών επιτοκίων. Η σχετική προσέγγιση βάση μοντέλων και ο στόχος είναι να μην υπάρχει η παραποίηση, η αλλίωση των μοντέλων ε, για να υπολογιστεί το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που διαρκώς πέφτουν τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό η Επιτροπή της Βασιλείας ε, εκπονεί προτάσεις για να βεβαιωθεί ότι αυτά τα εσωτερικά μοντέλα δεν αποτελούν αντικείμενο αλλοιώσεων και παραχαράξεων. Υπάρχει κάποια αναστάτωση λοιπόν. Βλέπουμε φόβος να επικρατεί με την αύξηση των κεφαλογικών απαιτήσεων που θα είναι σημαντικός και Ο Επίτροπο Ντομπρόφσκη μα είπε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ίσω να μην ε, εφαρμόσει αμέσω τι συστάσει τη Επιτροπή τη Βασιλεία. Εδώ λοιπόν εσεί τι βλέπετε. Βλέπετε να υπάρχει αυτή η αλλίωση των ιστορικών μοντέλων και επιτοκίων βάσει των αναγκών των ΜΕ και των ΔΕ. Και επειδή τουλάχιστον και τι Ολλανδικέ τράπεζε, ζητήσατε να υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά μόχλευση ε, προσωπικός. Πώς βλέπετε εσείς την αύξηση των κεφαλαχικών απαιτήσεων και την απειλή να μην προσπογράψουμε αμέσω τι απαιτήσει τη Επιτροπή τη Βασίλεια. Ε, κοιτάξτε, για τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα είναι ζωτική σημασία και για τους ίδιου τους πελάτες και για τους επενδυτές να μπορούν να εμπιστευτούν το προφίλ κινδύνου που τους ε, δίνει και τους περιγράφει η ίδια τράπεζα για τον εαυτό τη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν σαφή κριτήρια για να μπορεί να υπάρχει και αυτή η εμπιστοσύνη. Αυτή τη στιγμή συζήτηση γίνεται για τα εσωτερικά μοντέλα και όντω δεν είμαι κατά χρήση αυτών των εσωτερικών μοντέλων. Διότι λίγο πολύ λέμε ότι οι Αμερικανοί τα έχουν, α τα έχουμε κι εμεί. Οι Ευρωπαίοι λένε ότι ε, οι Αμερικανοί μάλλον λένε ότι δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα, εμεί λέμε ότι μπορούν να έχουν και κάποια αξία. Θα πρέπει απλώ να βεβαιωθούμε ότι η ποιότητα αυτών των εσωτερικών μοντέλων είναι περισσότερο προστατευμένη. Δηλαδή, Μπορεί να πρέπει να υπάρχει και ένα κατώτατο όριο για την ε, βαρύτητα των κινδύνων. Αυτή θα πρέπει να είναι η σωστή προσέγγιση, για να είμαστε απόλυτα βέβαιοι, και όχι επειδή απλώ μα το λένε οι Αμερικανοί, αλλά γιατί είναι προ το δικό μα όφελο να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία για την ποιότητα τη αξιολόγηση κινδύνου που προέρχεται από τα εσωτερικά μοντέλα και οι επόπτε μα να είναι σε θέση να ορίσουν την ποιότητα αυτών των εσωτερικών μοντέλων. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση για να προχωρήσουμε τώρα στι όλε τις διαπραγματεύσεις. Όντω υπάρχουν πολλές ε, διαμάχε, απειλέ για ε, διαφωνίες, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα Όμω, εν τέλει, αυτό που προέχει είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα. Και γι' αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε τα πρότυπα τη Επιτροπή τη Βασιλεία και να παραμείνουμε στο δυνατό πιο κοντά σε αυτά τα πρότυπα. Ε, το να αποκλίνουμε από αυτά θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση, την οποία θα, δεν θα προτιμούσα ω επιλογή. Αλλά α μην ε, προλαμβάνουμε τα συμπεράσματα. Η διαδικασία τη Βασιλεία δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κοινό έδαφο για να συμφωνήσουμε και να δούμε πώ θα προχωρήσουν τα εσωτερικά μοντέλα. Να υπάρχουν λοιπόν εσωτερικά μοντέλα αλλά και ε, πρότυπα ποιοτητα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η βαρύτητα του κινδύνου αντιμετωπίζεται με τρόπο σοβαρό και μπορούμε να δείξουμε εμπιστοσύνη. Έχετε προτείνει όμω και ανώτερο επίπεδο μόχλευση για τις τράπεζες. Και όχι μόνο για τη δική μα τη χώρα, αλλά και εκτό Ολλανδία. Θεωρώ λοιπόν από την απάντησή σας και συμπεραίνω ότι είστε υπέρ του να υπάρχει και ένα κατώτατο όριο για του κινδύνου. Το κατώτατο όριο για του κινδύνου μπορεί να είναι χρήσιμο όντω για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τα αποτελέσματα των ιστορικών μοντέλων. Τώρα για το ποσοστό μόχλευσης, όπω ξέρετε, Υπάρχουν ελάχιστε απαιτήσει 3% αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και αυτό δεν έχει οριστεί ω μόνιμο αναγκαστικά όριο για τι κεφαλαιοκέ απαιτήσει. Είναι μέρο ε, των διαπραγματεύσεων για, τους, για τις μεγάλες τράπεζες, συστημικά πιο εύστοχα, ε, πιο ενδιαφέρουσες. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να το δούμε ξανά αυτό το ποσοστό και πολλές φορές έχει υποθεί ότι αυτές οι τράπεζες έχουν πολλές πιστώσεις. Αυτό το έχουμε δει από την εμπειρία μας στην Ολλανδία. Έχει βελτιωθεί το κλίμα του προς τις τράπεζες, η χρηματοδότησή τους έχει αυξηθεί και το γεγονός ότι έχουν μεγαλύτερο ε, όγκο αξιοχρέων, αξιογράφων μάλλον, έχει ε, τονώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών για να αντιμετωπιστούν ίσως ε, και κάποια μελλοντικά προβλήματα. Όμως, ίσως αυτό είναι υπερβολικά τεχνικό για τις τωρινές μας ανάγκες αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν τα σωστά πρότυπα ποιότητα, το σωστό ποσοστό μόχλευση και κανένα από αυτά να μην γίνει δεσμευτικό στο όλο μοντέλο. Θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν. Είναι όμω ένα απαραίτητο στοιχείο τα κριτήρια ποιότητα ε, για την ε, μόχλευση του κινδύνου. Ευχαριστούμε. Στην Επιτροπή τη Βασιλείας θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία και να δούμε ποια θα είναι τα επιτόκια μόχλευσης στο πλαίσιο αυτό. Ο κύριος Χέης. Καλώς ήρθατε και πάλι κύριε Ντάισελμπλουμ. Πριν από λίγους μήνες ε, σας είχα ευχαριστήσει ε, για την έκθεση που πέρασε την περασμένη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο. Με την Ολλανδική Προεδρία είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ αγαστά και σας ευχαριστώ πολύ. Είπατε προηγουμένως ότι είστε καθολικός και εγώ καθολικός είμαι. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να κάνεις όρκο σιωπής ε, στην πολιτική. Και τώρα έχει πέσει μια ομερτά για το Brexit. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε. Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη χώρα μου και για τη δική σας χώρα, αλλά το λέω και ως ένας από τους 27, όχι ως Ιρλανδός βουλευτής. Ε, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κατακαιρματισμένε αγορές. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ αλληλένδετο σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά και στις κεφαλαίες Είναι πολύ σημαντικό για την Ένωση αυτό το κεφάλαιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και πραγματικά υπάρχει μια ανησυχία και σε σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένω ε, στον συνάδελφο Μάιερ, ότι οι εξωτερικοί κραδασμοί μπορεί να μα επηρεάσουν. Ε, και πώς λειτουργούν αυτές οι αγορές. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι ισχυρές αγορές, βαθύτερη εδραίωση και όχι κατακαιρματισμό και ε, πολυδιάσπαση. Ε, έχετε σκεφτεί, προβληματίζεστε αυτό τον καιρό ως πρόεδρος του Eurogroup για όλα αυτά τα θέματα. Ο Υφυπουργό ε, Οικονομικών στη Γερμανία είπε το εξή πολύ ενδιαφέρον. Για να μπορούν 27 στο μέλλον να έχουν καλέ σχέσει με τους Βρετανού, θα πρέπει οι Βρετανοί να δεχτούν τουλάχιστον όλες τις υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίε, τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς και σιωπηρά να αναγνωρίσουν για το μέλλον ότι αν θέλουμε να έχουμε σχέσει, θα πρέπει να το αναγνωρίσουν εκείνοι και να δέχονται και τους κανόνες των 27. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Αυτό μιλάει για ε, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, έτσι, όχι για την ελεύθερη κυκλοφορία. Ως πρόεδρος του Eurogroup, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε αρνητικό αντίκτυπο ε, ε, για τα δημόσια οικονομικά της Ευρωζώνης ως συνέπεια του Brexit. Είπατε ότι είναι στο 1,6 σταθμικά της 100 ή 1,7 η αύξηση του ΑΕΠ και είναι πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα έτη. Εντάξει, αλλά εγώ ανησυχώ κατά πόσο θα επηρεαστούν τα δημόσια οικονομικά της Ευρωζώνης από το Brexit και θα σας ήμουν ευγνώμων αν απαντούσατε. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω κάνει ορκοσιοποίηση για το θέμα του Brexit σε καμία περίπτωση και χαίρομαι που κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. για το χρηματοπιστωτικό τομέα, το να λέμε ότι προτιμότερο θα ήταν να δεχτούν απολύτως οι Βρετανοί όλες τις απαιτήσει και τα πρότυπα που έχουμε τώρα, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα εκτός Τραπεζικής Ένωσης που ήδη ε, υπάρχει πρόβλεψη απόκλησης από τις προδιαγραφές και τα πρότυπα. Το δεύτερο είναι πιο σημαντικό. Τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν μπορούν να πούν οι Βρετανοί ότι δεχόμαστε τώρα ε, το, την κοινή πολιτική και το βάζουμε στην ομοθεσία μας. Δεν λύνεται έτσι το θέμα. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε ε, σε μια τρίτη χώρα να έχει πλήρη πρόσβαση και ίδια δικαιώματα στη χρηματοπιστωτική αγορά χωρίς να σέβεται τα υπόλοιπα προστασία καταναλωτών, κεφαλαϊκές απαιτήσεις κλπ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ψάχνουν ένα νορβηγικό μοντέλο ε, για τις χρηματαγορές, ε, αλλά οι Βρετανοί ζήτησαν ε, το Brexit για λόγους κυριαρχίας. Δεν συνάδει με το νορβηγικό μοντέλο. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το κέντρο για τα χρηματοπιστωτικά και τα κεφαλαιακά της Ευρωζώνης να είναι εκτός Ευρωζώνης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει δικούς του κανόνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παρόλο που είμαι μέγας οπαδός των Βρετανών και οι Ολλανδοί ε, έχουμε μεγάλες σχέσεις ε, και εμπορικέ μαζί τους. Ε, νομίζω εσείς στη Ιρλανδία είστε η πρώτη χώρα και εμείς η δεύτερη στην Ολλανδία στι εμπορικέ μας σχέσεις. Ε, Παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε τι επίπτωση θα έχει αυτό στα οικονομικά. Το γεγονός και μόνο ότι μπαίνουμε σε μια φάση αστάθειας, αβεβαιότητας για τις μελλοντικέ σχέσεις θα επηρεάσει τις οικονομίες μας, κυρίως τη Βρετανική, διότι οι επενδυτές προστατεύουν τους κινδύνους που πρέπει να πάρουν. Παίρνουν αποφάσεις φέτος του χρόνου, ε, σε δύο χρόνια, δεν ξέρουν πού θα βρίσκεται η κατάσταση. Και ξανασκέφτονται πού θα επενδύσουν. Δεν χαίρομαι που το λέω αυτό. Αλλά αυτό θα αρχίσει να έχει αντίκτυπο και στο City και στη Βρετανική οικονομία του χρόνου και τα επόμενα έτη. Εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε όσο γίνεται και να είμαστε έτοιμοι όσο και εκείνοι, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα αρνητικά, γιατί δεν είναι δικό μας συμφέρον να βλαφθεί η ε, Βρετανική οικονομία ή να αφήσουμε τις δικές μας οικονομίες να υποστούν ζημία. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αλλά θα είναι δύσκολη περίοδος, ιδιαίτερα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Σίλβα Περέιρα. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε πολύ για τις ε, ανακοινώσεις της Επιτροπής. Ήταν θετική η στάση που εκφράστηκε για τις χώρες της Ευρωζώνης και σημειώνουμε ότι το Eurogroup βεβαίως θα συζητήσει περαιτέρω για την ε, ανακοίνωση αυτή. Επίσης, να σημειώνω ότι αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι πέραν του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, ευθύνεται στα κράτη-μέλη το τι θα κάνουν και η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι πρόκειται για σύσταση που δεν είναι δεσμευτική. Επιπλέον λέτε ότι αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης η πρώτη αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να βεβαιωθεί για την εφαρμογή του συμφώνου. Δεν νομίζω ότι διευκολύνει τίποτα να παραγνωρίζουμε το θεμελιώδες ζήτημα που αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί επιτάπητος. Η όλη συζήτηση δεν έχει να κάνει με την εφαρμογή του συμφώνου ακριβώς. Η Επιτροπή δεν μιλά, ούτε σχολιάζεται με συμμόρφωση με το σύμφωνο. Η όλη συζήτηση γίνεται για το κατά πόσον είναι ορθή, εσφαλμένη δημοσιονομική πολιτική. Και το όντι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θε, αμφισβητεί την ε, δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Η Επιτροπή λέει, και εδώ ανοίγω το παράθεμα, βάσει των τελευταίων οικονομικών και δημοσιονομικών στοιχείων, η πλήρης επίτευξη των απαιτήσεων των δημοσιονομικών όπως περιέχονται στις αναχώρασεις τάσεις του Συμβουλίου που τον Ιούλιο μόλις πριν τέσσερις μήνες ε, υπόθηκαν θα οδηγήσει ε, κατά συνάθρηση σε ε, περιορισμένη κατά μέσο όρο δημοσιονομική στάση για το 2017 και 2018 ενώ η οικονομική κατάσταση ζητά ε, να είμαστε επεκτατικοί στη δημοσιονομική μας πολιτική. Άρα, αυτό σημαίνει ότι οι τάσεις αναχώρα απαιτούν περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, όμως οι οικονομικές καταστάσεις, η οικονομική πραγματικότητα απαιτούν το αντίθετο. Οπότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά αμφισβητεί. Αμφισβητεί τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Συμφωνώ λοιπόν όταν λέτε ότι πρέπει να φουγκραστούμε και τα κρατημέλη, να δούμε τι θα μας πούνε. Εντάξει, αλλά υπάρχει μια αξιολόγηση που πρέπει να κάνει και το Eurogroup από μόνο του. Δεν μπορούμε διαρκώς να βάλουμε την όλη υπόθεση. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την ανάγκη να υπάρχει μια μετριοπαθώς επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Νομίζω το πραγματικό ερώτημα είναι στις χώρες που υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις θέλουν να το κάνουν Νομίζω κάποιες δεν υποχρεωθούν, διότι το πλεόνασμα ε, είτε έχει ανακοπεί είτε έχει φτάσει. Δηλαδή έχουν φτάσει σε ψηλά επίπεδα και πλησιάζουν την πλήρη απασχόληση. Ενώ σε άλλες χώρες υπάρχει υψηλή ανεργία και μεγάλη διαφορά ως προς το πλεόνασμα με τις πρώτες, οπότε δεν υπάρχει και περιθώριο για επενδύσεις. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο του οικονομικού κύκλου και αυτό είναι μείζωνα πρόκληση. Δεν ξέρω μπορεί να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό η όλη αντίληψη της δημοσιονομικής τάσης της Ευρωζώνης είναι τόσο περίπλοκη. Ναι, μπορείτε εν γέννη να πείτε ότι υπάρχει μια μετριοπαθώς ε, επεκτατική πολιτική για την Ευρωζώνη. Θα έπρεπε μάλλον να υπάρχει. Αλλά πώς αυτό θα επηρεάσει την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Η Επιτροπή δεν έχει δώσει εδώ απάντηση. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φαντακίντελαρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Ε, στο δελτίο ενημέρωση που ετοιμάστηκε για αυτή τη συζήτηση, εκεί υπογραμμίζεται για μας ότι οι συζητήσεις θεματικές δεν είναι αποτελεσματικές και μπορούν να βοηθήσουν στο να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Και ρωτώ, εσείς ε, συμφωνείτε με αυτό και αν ναι, μπορούμε να βελτιωθούμε περαιτέρω. Το δεύτερο, πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, το Eurogroup είχε θεματικές συζητήσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ρωτώ, πιστεύετε ότι υπήρξε ουσιαστική βελτίωση στα κράτη-μέλη και αν ναι, την πρόσφατη πρόταση σχετικά με την οδηγία για την αναδιάρθρωση ε, της, ε, του πλαισίου μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τι είπατε στην αρχή, το κατάλαβα καλά. Είναι ένα έγγραφο από τους Έντερλαν και Χάσ. Αυτό ε, χρησιμοποιήθηκε ως ενημερωτικό δελτίο για το διάλογο. Και εκεί αναφέρεται ότι οι θεματικές συζητήσεις που γίνονται στο Eurogroup είναι αναποτελεσματικές. Δεν ξέρω, ε, δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω διαπιστώσει ότι αξιολογούνται οι θεματικές συζητήσεις στο Eurogroup. Άρχισα να το διαβάζω κι εγώ, θα το δω, να δω. Αυτό που έχει σημασία είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρωζώνη. Γιατί εδώ υπάρχει δυνατότητα για τα κρατημέλη, για μεμονωμένους θεσμούς, για τράπεζες να αναλάβουν την ευθύνη, για επόπτες, για την ΕΚΤ, για την Επιτροπή και έγιναν αρκετές συζητήσεις στο Eurogroup όλα αυτά να τα συνενώσουμε Είχαμε μία συζήτηση με τον Ντανιέλ Νουή από το SSM που ελέγχουν, εποπτεύουν ε, τις δικές μας τις τράπεζες. Να δούμε αυτοί πώς αντιμετωπίζουν το θέμα. Πώς ε, θα πρέπει μία τράπεζα να αναδιαρθρώνεται ε, και αυτό το θέμα το συνδυάσαμε με αυτά που μπορούμε να κάνουμε και εμείς ως εθνικοί νομοθέτες για τα πλαίσια ε, πτώχευσης. Ξέρετε ότι τα πλαίσια και τα όρια πτώχευσης ε, διαφέρουν πάρα πολύ στα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν έχουμε καταρτήσει μια σειρά προδιαγραφών ε, για το πόσο καιρό χρειάζεται παραδείγματος χάρη για να περάσει κανείς μέσα από μια διαδικασία πτώχευσης σε ορισμένες χώρες 1,5 μέχρι 2 χρόνια, σε άλλες πάλι 7 μέχρι 8 χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιες ε, διαφορές σε εθνικό επίπεδο. Κατόπιν ως Επιτροπή καταθέσαμε μία πρόταση για να γίνει κάποια δουλειά είτε για την εναρμόνιση αυτών των ε, ορίων ή να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό όριο και ένα πλαίσιο για το τι πρέπει να γίνει σχετικά με το πλαίσιο αναδιάρθρωσης που ε, θα επιτρέπει την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση που είχαμε στο Eurogroup ε, με τους διάφορους θεσμούς και τις εθνικές κυβερνήσεις, αυτή η συζήτηση δημιούργησε μια νέα δυναμική και πάρα πολλοί είπαν ε, ξεχάστε το θέμα των πτωχεύσεων, είναι πάρα πολύ περίπλοκο και δεν θα υπάρξει καμία εξέλιξη. Δεν πάει έτσι όμως, είναι καθοριστική σημασία σε αυτό το θέμα οι πτωχεύσεις και είναι σημαντικό για να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη νέων επονδετών στην Ευρωζώνη. Αυτοί πρέπει να ξέρουν πώς λειτουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι πτωχεύσεις, αν είναι αποτελεσματική διαδικασία, αν μπορεί κανείς να πάρει πίσω τα λεφτά του, αν όλα πάνε στραβά, ε, τι γίνεται με τις εθνικές κυβερνήσεις, ε, με την Κομισιόν. Ε, αυτά όλα αποδεικνύουν ότι η δική μας προσέγγιση είναι σωστή. Alfred Sand. Ευχαριστώ τα τελευταία χρόνια. Ε, φαίνεται να υπάρχει διάθεση να πλήσει το χάσμα μεταξύ των χωρών που τα έχουν καταφέρει και αυτών που τα καταφέρνουν, αλλά αυτό αυξάνεται. Λέμε ότι θέλουμε μηδενική φτώχεια και ανεργία σε κάποιε χώρε ενώ σε άλλε βλέπουμε διαρκώ να είναι εξαρτημένε από το χρέο, να υπάρχει υψηλή ανεργία, να υποχωρεί το κράτο πρόνοια και να αυξάνεται η φτώχεια. Αυτό ε, παρατηρείται σε κράτη τη Ευρωζώνη και μη. Απλώ κάποιοι είναι δεσμευμένοι από τι κανόνες τη νομισματικής και οικονομικής ένωσης. Με την ε, τη έκθεση ανάπτυξη του 2017 ζητήθηκαν για βήματα πρόοδου από την Επιτροπή. Λέγεται ότι κάποιε χώρε θα πρέπει να αξιοποιήσουν το δημοσιονομικό του περιθώριο για να περάσουν σε επενδύσει ακόμη και διασυνοριακέ. Ακούσαμε τα σχόλιά σα, αλλά ω πρόεδρο του Eurogroup και του επερχόμενου, το Δεκέμβριο. Πόσο πιθανό θεωρείτε τα κάτι μέλη τη Ευρωζώνη να μην συμφωνήσουν με την Επιτροπή. Υπάρχουν κάτι μέλη που μπορούν να εφαρμόσουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, έχοντα υπόψη το τωρινό πλαίσιο κανόνων. Γιατί και ο ΣΑ μόλι χθε σύστησε να γίνουν περισσότερε επενδύσει. Ω πρόεδρο του Eurogroup, Θεωρείτε ότι οι συστάσεις ε, θα έπρεπε να εφαρμόζονται καλύτερα. right. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η διαδικασία σύγκλησης τελικά κατέντησε να είναι διαδικασία απόκλησης. Και αυτό είναι μια απειλή κατά της κοινότητάς μας, της νομισματικής μας ένωσης, παρόλο που προσφάτως αντεστράφει, Εάν δείτε τα ποσοστά ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αυτό το διάστημα, θα δείτε ότι η διαδικασία ήδη ε, έχει αρχίσει να μεταβάλλεται και να αντιστρέφεται. Τα ποσοστά ανάπτυξη σε κάποιε από τι χώρε που είχαν προβλήματα προηγουμένω τώρα έχουν αυξηθεί πολύ. Στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο. Η οικονομική ανάπτυξη ανάκαμψη είναι μια πραγματικότητα. Και είναι και μεγαλύτερα τα ποσοστά από ό,τι στι χώρε που τα πηγαίνουν έτσι κι καλά. Χρειάζονται περαιτέρω βήματα ω προ τι μεταρρυθμίσει μετά τι αναχώρασει τάση. Βεβαίω, συμφωνώ. Αλλά η μείζων πρόκληση για του πολιτικού ευθύνοντε είναι η εξή. Όλοι έχουμε πιεστεί. Γι' αυτό κοιτάζουμε τόσο πολύ τα αποτελέσματα και το να είμαστε αποδοτικοί σε ό,τι κάνουμε για να δώσουμε νέες ευκαιρίες στον κόσμο, τώρα που αρχίζουμε να βγαίνουμε από την κρίση. Δύσκολη στιγμή, διότι ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα και είναι αργή η διέξοδος από την κρίση. Όμω θα αρχίσουν να φέρονται τα πρώτα σημάδια τη σύγκριση. Υπάρχουν ενδιαφέρουσε διαφορέ ε, στα ποσοστά ανάπτυξη και τη δυναμική τη στι διάφορε χώρε τη Ευρωζώνη αλλά να πω ότι Κάποιε χώρε θα πρέπει να αυξήσουν τα ποσοστά ανάπτυξή του, ακόμη και αν δεν το σκεφτόμαστε. 1% για τα μεγάλα κράτη τη Ευρωζώνη δεν είναι αρκετά καλό ποσοστό. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώσαμε αυτή μα τη συζήτηση και τον ολοδιάλογο. Εντατικό. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ, Γερούν, που ήσουν εδώ και πραγματικά ανυπομονούμε για τη συζήτηση στο Eurogroup για τα θέματα αυτά. Και ελπίζω να υπάρξει επικοδομητική προσέγγιση. και να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ του τωρινού νομοθετικού πλαισίου και των κυριάρχων δικαιωμάτων των εθνικών κρατών μελών, αλλά και των όσων ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας και εκείνη που παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων και το τι θα συμβεί στο σύνολο της Ευρωζώνης και το πώς τη μεταχειρίζεται. Οι συστάσεις πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμόζονται. Η όλη συζήτηση λοιπόν ε, είναι και συζήτηση ουσίας για το πώς το πολιτικό μείγμα μπορεί να αποτελέσει πραγματικά ε, κάτι το θετικό για την πραγματική οικονομία. Επίσης ελπίζουμε να επιτελεστεί πρόοδος για την Ελλάδα και να προχωρήσουμε σε μια επικοδομητική κίνηση και εκεί. Σας ευχαριστώ. και ελπίζω να ξανάρθετε σύντομα για να συνεχίσουμε το διάλογό μας. Ευχαριστώ.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 Να περάσουμε τώρα στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, ε, δηλαδή το, τη χρονοθυρίδα για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και τα εκτελεστικά μέτρα. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο PSD2 και συγκεκριμένα το RTS για τη διαπίστωση των στοιχείων των ε, πελατών και καταναλωτών και ε, την ε, και την διαπίστωση της ταυτότητας. μετά την πρώτη συζήτηση τον Απρίλιο θα συζητήσουμε το σχέδιο των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την ασφαλή επικοινωνία, διότι αυτή τη στιγμή Η EBS σε συνεργασία με την ECB ετοιμάζουν ένα βελτιωμένο RTS ώστε να υπάρχουν εύρωστα μέτρα βάσει του ETS 2 και η EBA έχει ασχοληθεί με το σχέδιο του RTS, e το οποίο το είδαμε από τον Οκτώβριο, αλλά έχουμε πολλά σχόλια και απαντήσεις. Και εδώ θα χρειαστεί να διευκρινιστούν κάποιες από τις αρχές που διέπουν το RTS2 για τους παρόχους και τους καταναλωτές. για τις υπηρεσίες πληρωμών και τις, ε, τους κανόνες που διέπουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στις 24 Οκτωβρίου σχολιάσαμε με επιστολή μας στην EBA το RTS και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι μια καλή αφορμή για να δούμε πώς θα χειριστούμε το όλο, ε, τον όλο φάκελο. Είναι σημαντική και τεχνολογική ουδετερότητα, αλλά και κάποιες εγγυήσεις οι οποίες πρέπει να προκύψουν από το άρθρο 63 εδάφιο 3 ως προς τις εγγυήσεις και την ταυτοποίηση και ένα πολύ σημαντικό σημείο για τις εξαιρέσεις. και τη δυνατότητα να προβλεφθεί περισσότερη ευελιξία. Έχουμε σημαντικά ζητήματα να συζητήσουμε Να χαιρετήσω τον κύριο Σάλε, τον Γενικό Διευθυντή Φίσμα από της Γενική Διεύθυνσης από την και τον πρόεδρο της CBA, τον κύριο Ερία, καθώς ε, και από την Γενική Διεύθυνση Τάξη τον Γενικό Διευθυντή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την διπλωματική μας ομάδα. Να ξεκινήσω δίνοντα το λόγο στην EBA πρώτα. Ο κύριος Ενρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που κάλεσα την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Έχετε την ευκαιρία, μας δίνετε μάλλον την ευκαιρία ε, να σας παρουσιάσουμε την τελευταία ε, εργασία μας, το τελευταίο διάστημα. Ε, έχουμε στόχο τη σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βάση καταστατικού ε, και ε, μεγαλύτερη ε, δυνατότητα ανταγωνισμού για τις πληρωμές, μια λύση φιλική προς τον καταναλωτή και να υπάρχουν αγορές, μια πανευρωπαϊκή αγορά. Σε τέσσερα από τα θέματα αυτά έχουμε εκδώσει ήδη κάποιες προτάσεις. Μέχρι τον επόμενο Φεβρουάριο θα ακολουθήσουν και άλλα δύο. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την ταχύτητα. Έχουμε προβλήματα και οικονομικών πόρων και ανθρωπίνων πόρων. Πάντως, κατά τη διάρκεια της εντολής μας, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές, διόρτιες, ε, για την κοινή ε, προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή από κοινού διαχειρίζονται αυτό ε, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, ανταγωνιστική ζήτηση. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται ε, στις αγορές ε, στην ενιαία αγορά πληρωμών. Είναι πολύ διαφορετικές οι ε, προδιαγραφές για το ERTS και ε, υπάρχει ενδεχομένω και γεωγραφικός κίνδυνος. Επίσης θα πρέπει να είμαστε προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των καταναλωτών και η παρέμβαση στις πληρωμές να είναι όσο γίνεται χαμηλότερη και να είναι το περιβάλλον φιλικό όχι μόνο προς τους χρήστες ε, αλλά και τα τρίτα μέρη για να γίνονται απρόσκοπτα οι συναλλαγές. Ποια είναι τα προβλήματα ε, και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και πώς τα αντιμετωπίσαμε, θα ήθελα λίγο να σας αναλύσω και στην επιστολή Φέρμπερ και Ταγιάννη που έλαβα τον Οκτώβριο ε, εξ ονόματος της ε, Διαπραγματευτικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για το PSD2 και να σας πω και ποια είναι τα βήματα που απομένουν. Πρώτον, για τη διαδικασία που έχουμε καλύψει. Το RTS είναι βασικό στοιχείο για τους στόχους PSD2, για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη διευκόλυνση καινοτομία και τις ασφαλείς πληρωμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές, τις προκλήσεις, ε, όπως είναι οι πληροφορίε για το λογαριασμό και ε, τη διαδικασία πληρωμών. Κυρίως οι Τράπεζε τα χειρίζονται αυτά για την πρόσβαση στους λογαριασμούς πληρωμών. 12 μήνες μόνο είχαμε για να ε, κάνουμε αυτή την εργασία. Το θέμα είναι πολύ περίπλοκο και πολύ δύσκολο από την αρχή καταλάβαμε ε, και ήταν ξεκάθαρο ότι θέλαμε καθοδήγηση και βοήθεια. Γι' αυτό πονήσαμε ένα έγγραφο συζητήσεων και, στις, και λάβαμε 118 παρακαλώ ε, απαντήσεις από ενεχομένους της αγοράς και άλλους ενδιαφερομένους. Αξιολογήσαμε αυτές τις απαντήσεις ε, και οι τράπεζες και οι τρίτοι ε, πάροχοι εκλήθησαν να συζητήσουν και στη συνέχεια ακολούθησε ένα έγγραφο διαβούλευσης το οποίο δημοσιεύσαμε τον Αύγουστο του 2016. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έκανε 20 διαφορετικές διασκέψεις παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρουσιάσει τις σκέψεις της να γνωρίζει ακόμα και πιο μικρή ε, ε, νεοφυής επιχείρηση ή μικρομεσαία τις δυνατότητες που έχει για το RTS έτσι ώστε να υπάρχει ε, σωστή ισορροπία. Ε, με επιτυχία αυτές οι προσπάθειές μας. 226 απαντήσεις λάβαμε στο έγγραφο διαβούλευσης, πάνω από 2.000 σελίδες συνολικά. Ε, και αυτό νέο ρεκόρ για τη διαβούλευσή μας. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το RTS και γενικότερα πόσο συνεισφέρουν ε, οι διάφορες πλευρές. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο προχωρήσαμε στην αξιολόγηση και περίπου βρήκαμε 260 διαφορετικές ε, ανησυχίες ή αιτήματα διευκρινήσεων αξιολογήσουμε και θα κοιτάξουμε αν θα απαντήσουμε και με ποιο τρόπο στο έγγραφο αυτό. Και τέλος ε, θα υπάρξει ένας πίνακας για feedback ε, που θα απαντούμε σε όλους όσους ε, μας υπέβαλαν τις προτάσεις τους. Στον πίνακα συνοψίζουμε τις 260 ανησυχίες και αιτήματα και εξηγούμε γιατί προχωρήσαμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι Μέγα αριθμό των ετοιμάτων δεν συνδέονται με το RDS αλλά με το ίδιο PSD2 και πώς ερμηνεύονται οι διατάξει. Αυτά δεν είναι θέματα τη Ευρωπαϊκή Τραπεζικής Αρχής. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα συζητούμε με ποιο τρόπο θα γίνεται η επικοινωνία. Εμεί λοιπόν δεν λειτουργούμε απομονωμένοι, γι' αυτό σα τα λέω αυτά, δεν ζούμε σε κανένα ε, ε, πύργο φιλντισένιο, αλλά συνεργαζόμαστε με την κοινωνία και με τους ενδιαφερόμενους φορείς με πλήρη διαφάνεια. Θα ήθελα τώρα να αφαιρθώ σε τρία βασικά αιτήματα από τα 260 που μας ανέφεραν πολλοί και επίσης οι βουλευτές Φέρμπερ και Ταγιάννη στην επιστολή τους. Αυτά είναι τα όρια, τα νομισματικά, η διαδραστική επικοινωνία ε, που η επιστολή τώρα φέρει ως άμεση πρόσβαση και κάποιες εξαιρέσεις. Ε, ποια είναι τα νομισματικά όρια, το κατόφλι δηλαδή. Προβλέπεται στο σχέδιο για πληρωμές εξ αποστάσεως ένα κατόφλι 10 ευρώ. Ορισμένοι λένε ότι εδώ έχουμε ε, λίγες πληρωμές που είναι κάτω των 10 ευρώ, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ε, και δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει αυτός... στους καταναλωτές και στις εταιρείε. Οι ανέπαφες ε, συναλλαγές και οι εξαποστάσεως ε, έχουν υψηλότερο κίνδυνο απάτης. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δημιουργήσουμε τρόπους πληρωμής φιλικούς προς το χρήστη και όσο και ασφαλής. Έχουμε λάβει πολλά σχόλια και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξισορροπήσουμε εκεί ε, την ε, άνεση και τη βολική χρήση για τους καταναλωτές με την ε, ασφάλεια και την προστασία των συναλλαγών. Άλλο πρόβλημα είναι η επικοινωνία, η άμεση πρόσβαση και πώς χρησιμοποιείται το σύστημα αυτό για να υπάρχει πρόσβαση σε ένα λογαριασμό πληρωμών. Αυτή είναι η λεγόμενη άμεση πρόσβαση ε, μέσω από μια διαδραστική επιφάνεια τράπεζας και ε, πελάτη για online banking. Αυτές ε, οι διαδικασίες προβλέπονται στο άρθρο 66.4 και 67.3 του PSD2 σε σχέση με τη μη διάκριση και τη διάδοση της πληροφορίας. Απαντώντας στις δύο πρώτες αιτήσει, τα αιτήματα μάλλον, θα πρέπει να δούμε πώς ορίζεται η εντολή μας στο αρθρο 91 1 91.1d, από το οποίο δεν μπορούμε να αποκλίνουμε ως τραπεζική αρχή. Τι ορίζεται εκεί, ότι η EBA θα ορίσει τις απαιτήσει για κοινή ε, ανοιχτή και ασφαλή επικοινωνία για ενημέρωση, ταυτοποίηση, ε, πληροφόρηση καθώς και την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας. Άρα στην εντολή μας δεν έχουμε ως στόχο να διευκρινίσουμε τα RTS ή το PSD2. Αυτό που αναφέρεται στην επιστολή σας ως direct access, άμεση πρόσβαση. Ε, μόνο στο ε, Τελογική Σκέψη 32 υπάρχει μια αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η, πρόταση, η πρόσβαση. Αλλά δεν είναι ε, κεκτημένο δικαίωμα. Από την άλλη, ούτε οι αιτιολογικές σκέψεις, ούτε τα άρθρα ε, ορίζουν την άμεση ε, πρόσβαση. Ή ότι το, το scraping μπορεί να είναι μια παραλλαγή. Ε, Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι σημαίνει λοιπόν άμεση πρόσβαση, ακόμα και αν ήταν στην εντολή μας να το ζητούμε. το σχέδιο RTS που προτείνουμε λοιπόν, ε, δεν αναφέρει καθόλου την άμεση ή την έμεση πρόσβαση όπως η οδηγία ίδια. Αντίθετα, το άρθρο 19 του σχεδίου ΕΡΤΕ ζητάει ότι ε, Όταν υπάρχει μια δυνατότητα επιγραμμική πληρωμή, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια διαδραστική επιφάνεια πληροφορία. Αυτό δεν ε, συγκεκριμενοποιεί αν θα είναι στην ίδια επιφάνεια με του εκείνη που χρησιμοποιούν οι πελάτες ή αν είναι μια ειδική επιφάνεια για τις τρίτες, τους τρίτους που θέλουν να έχουν πρόσβαση ε, στο λογαριασμό και σε πληροφορίες. Ε, αυτά δεν τα αναφέρει ούτε το RTS ούτε το PSD2 και θα μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι λένε οι ευρωβουλευτές. Για τη δεύτερη πρόταση, το RTS Επίσης ε, δεν συμπεριλαμβάνει τέτοια ε, διαταξίες και μένα γιατί περιλαμβάνεται στο άρθρο 97.5 του PSD2 και δεν θα υπήρχε λόγος ε, μια τεχνική προδιαγραφή να επαναλαμβάνεται σε άλλη νομοθεσία. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με τις εξαιρέσεις που έχουμε ως εντολή να Ε, δούμε που δεν ε, χρειάζεται για την πληρωμή ε, αυστηρή ταυτοποίηση του πελάτη. Είναι το κείμενο του πρώτου επίπεδου. Οι εξαιρέσει ορίζονται με την πολύ στενή έννοια και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάλυση με βάση το κίνδυνο. Για να δούμε, για να καταλάβουμε τι κρύβεται από πίσω, ποιο είναι το σκεπτικό. Γιατί η εντολή στο άρθρο 91, 97.1 συγγνώμη, προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα εξασφαλίσουν ότι ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμής ε, ε, ζητάει ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν γίνεται επιγραμμικά ε, η πληρωμή, όταν αρχίζει ηλεκτρονικά ή μέσω ενός διάβλου που υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης ή απάτης. Ο πρόεδρος τελειώνεται. Ναι, αυτή η μεσω ενος διαβλου που υπαρχει κινδυνος καταχρησης η απατης προεδρος τελειωνεται ναι αυτη η εξαιρεση δεν μπορεί να αποκλείσει ε, την, ε, το SCA το, την ισχυρή ταυτοποίηση του ε, πελάτη και υπάρχει κίνδυνο ο κανόνας να γίνει εξαίρεση. Η ε, πρόταση RTS δεν αναφέρεται σε αυτή την ανάλυση κινδύνου, ε, αλλά δεν σημαίνει ότι και την απαγορεύει. Άρα ε, τους παρόχους ε, υπηρεσιών πληρωμών να το συμπεριλάβουν αυτό σε επιπλέον μέτρο για τη μείωση της απάτης. Δηλαδή αυτά τα βλέπουμε εμείς ως συμπληρωματικά και όχι υποκατάστατα. Τώρα, συμπέρασμα. Τώρα να θεωρούμε όλα τα σχόλια από το έγγραφο της διαβούλευσης. Είμαστε βεβαίως στη διάθεσή σας ε, να μελετήσουμε σε βάθος τις ανησυχίες και ε, τα αιτήματα που διατυπώνονται και μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και είμαστε βέβαιοι ότι θα βρούμε τη χρυσή τομή. Ε, περιμένετε τον Ιανουάριο να σας παραδώσουμε την εντολή. Αρχές Φεβρουαρίου ε, και ελπίζουμε, θα είμαστε έτοιμοι να μην διακυβευτεί ο στόχος της εφαρμογής της οδηγίας το 2018. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πιερ εκτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μας για την ευκαιρία που μας δίνεται να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήθελα στην ε, παρέμβασή μου να επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα τα οποία θεωρώ είναι σημαντικά στο στην επιστολή της διαπραγματευτικής ομάδα του Ευρωκοινοβούλιο. Το πρώτο έχει να κάνει με την απευθείας πρόσβαση και το άλλο με την ανάλυση κινδύνου των ε, δοσοληψιών, των συναλλαγών. Πρώτα απ' όλα για την άμεση πρόσβαση. Δεν είναι καινοτομία του PSD2 ότι θα προβλέψει. Μάλλον είναι καινοτομία βήμα για το PSD2 ότι θα προβλέψει την πρόσβαση στις τράπεζες για τις ε, επιγραμμικές πληρωμές και το σύνολο των λογαριασμών. Εδώ έχουμε υποστήριξη στην πρωτοβουλία αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή αυτό θα ε, ενσωματωθεί πλέον στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι τράπεζες βεβαίως ε, αντιτάχθησαν. Όμως θα προχωρήσουν τα πράγματα και αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε λόγο να μην και οι ίδιες οι τράπεζες δεν βλέπουν τον λόγο να μην ε, μπορούν να προχωρήσουν σε έλεγχο των ε, πληρωμών των πελατών τους και των επιγραμμικών πληρωμών. Όλα αυτά τα λέω διότι θεωρώ ότι η σχέση μεταξύ τραπεζών και εξωτραπεζιτών στο θέμα αυτό έχει τελικά οδηγηθεί σε σύγκληση. Το PSD2 έχει καταλήξει σε ε, κοινά πρότυπα για τα θέματα αυτά και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την EBA για να το πετύχουμε αυτό, την αρχή των τραπεζών. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει συνένεση στην αγορά Οπότε, μάλλον χρειάζεται να ε, δημιουργηθεί μία, ε, μία πλατφόρμα η οποία να είναι τυποποιημένη. Και από την πλευρά των τραπεζών έχει εκφραστεί αυτή η ανάγκη. Αυτή η τυποποιημένη λοιπόν διεπαφή θα μπορούσε να λειτουργεί αποτελεσματικά, να είναι διαθέσιμη διαρκώς και να υπάρχουν και κάποιες ε, διευθετήσεις και λύσεις για την αντιμετώπιση κατεπηγόντων σε περίπτωση που δεν λειτουργεί. Η δική μας αρμοδιότητα θα είναι στο μέλλον να ορίσουμε τις απαιτήσει που αυτή η τυποποιημένη διεπαφή θα πρέπει να μπορεί να φέρνει εις πέρας και προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα. Αυτή την ανάγκη την έχουν εκφράσει κάποιοι από τους ενδιαφερομένους στην πράξη και το είπατε και εσείς στην επιστολή σας. Η απευθείας πρόσβαση, η οποία σήμερα προβλέπεται, θα πρέπει να διατηρηθεί εφόσον η τυποποιημένη διεπαφή δεν λειτουργεί εύρυθμα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το σκέλος να το καλύψουμε παρκώς και αποτελεσματικός και να εντοπίσουμε στο σχέδιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών τι σωστέ απαιτήσει ώστε η επαφή να λειτουργεί σωστά. Ε, μαζί λοιπόν φροντίζουμε με την EPA να εκπονήσουμε τις σωστές προτάσεις. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Ορισμένοι φοβούνται ότι όχι απλώς μπορεί να με λειτουργήσει αυτή η επαφή, αλλά ότι η e TPP δεν θα έχει πλέον πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που έχει σήμερα με τον τρόπο που λειτουργεί. Δηλαδή τις ίδιες με αυτές που έχει ο, ο πληρώνων στο τραπεζικό του περιβάλλον online. Άρα το πρόβλημα δεν είναι απλώς να γίνεται κουβέντα για το όλο θέμα, αλλά για το τι είδους πληροφορίες θα ανταλλάσσονται. Δεύτερο λοιπόν καθήκον θα είναι να εντοπιστούν οι κατάλληλες απαιτήσει για την ανταλλαγή πληροφοριών. Είπα τι πρέπει να κάνουν οι ρυθμιστές. Υπάρχουν όμως και αυτά που να κάνει η αγορά κατά την άποψή μας. Θεωρούμε ότι πέραν της οδηγίας αυτή και του σχεδίου για το RTS, ένα ε, σχετικό επίπεδο για τυποποίηση της αγοράς χρειάζεται προκειμένου να αναπτυχθεί ή να ε, καλλιεργηθεί η ανάπτυξη ανταγωνιστικής πανα, πανευρωπαϊκής ε, διευθέτησης των επιγραμμικών πληρωμών. Έχουμε συζητήσει εδώ με όλους τους αντιφερομένους φορείς, ακόμη και με αυτούς που έχουν εκφράσει ανησυχίες και ενδιασμούς προέκυψε συμφωνία με αυτή την ευκαιρία για την ανάγκη τεχνικών προδιαγραφών όπως η τυποποιημένη διαπαφή αλλά και λειτουργικά επιχειρησιακά ζητήματα για τα οποία η αγορά θα πρέπει να βρει κοινέ λύσεις εάν θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Το Συμβούλιο για τις Ελληνικές Υπηρεσίες του Ευρώ το οποίο ε, εκφράζει για τις ανάγκες ε, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εδώ, άρχισε από την Παρασκευή να κινείται προς την εξέβρεση αυτών των κοινών λύσεων. Με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων, ακόμα και αυτών που έχουν εκφράσει ανησυχίες. Για το δεύτερο θέμα, για την ανάλυση κινδύνων στις συναλλαγές, προτείνουμε τις εξής κατευθυντήριες γραμμές Πρώτον, τρία θα στοιχεία. Πρώτον, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η PSD2 θα αποτελέσει ένα άλμα ποσοτικό για τα στοιχεία των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ο νέος κανόνας είναι η αυστηρή ταυτοποίηση και επ' αυτού ο Ευρωπαίος νομοθέτης πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί πλήρη ασφάλεια των συναλλαγών. Δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσει. Δηλαδή ανάλυση κινδύνου για τι συναλλαγέ, ειδικά. Και τρίτη παρατήρηση, οι ανάγκε τη αγορά λαμβάνονται υπόψη πολύ σοβαρά προκειμένου να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να συνδυάσουμε τι ανάγκε αυτέ με τις απαιτήσει της οδηγίας πίστη 2. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Σάλλας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα συνάδελφοι. Έχουν ήδη λεχθεί πάρα πολλά από τους προλαλήσαντες και θα ήθελα να περιορίσω λιγάκι την ομιλία μου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ καλό ότι συλλογικά έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για αυτές τις ε, προδιαγραφές. Θα ήθελα λιγάκι να σας υπενθυμίσω γιατί συζητάμε όλα αυτά σήμερα να επανέλθω στις βασικές αρχές της Οδηγίας Υπηρεσιών Πλειονομών την υπαριθμών 2 ε, που πολλοί παίκτε σε πολλές χώρες θεωρούν ότι αυτή είναι μια πολύ καλή οδηγία. Γιατί ε, είναι καινοτόμα και βοηθάει ε, στο να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια πληρωμών. Επίσης, ωφελεί τους ε, καταναλωτές και τέλος, διότι φέρει σταθερότητα και ασφάλεια σε όσους συμμετέχουν στην αγορά. Γι' αυτό λοιπόν ας μην ξεχνάμε ότι ο αρχικός στόχος ήταν ότι είναι απαραίτητη αυτή η οδηγία και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους συνομοθέτες της Τώρα, όσον υπάρχει το πλαίσιο, το επίπεδο υπαριθμών 2, Ένα σημαντικό παράγοντα είναι η ασφάλεια. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε γιατί ε, έχει εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα. Η μεγαλύτερη ασφάλεια πληρωμών ήταν ένα σημαντικό αίτημα από τους επόπτες αλλά και από τις τράπεζες σε μεγάλο βαθμό για να γίνει ε, αποδεκτό, το ανοίγει η αγορά για νέους παίκτες και για τη FinTech. Επίσης, ε, σημαντικό ήταν να προσφέρεται ασφάλεια στους καταναλωτές όταν θέλουν ε, συναλλαγές διαδικτυακά, επιγραμμικά. Υπήρχαν πάρα πολλές απάτες και θέλω να σας υπογραμμίσω ότι σήμερα ε, το θέμα αυτό εξακολουθεί να παραμένει. Δεν θέλω τώρα να σας ε, βομβαρδίσω με στατιστικά δεδομένα, αλλά είναι σαφές ότι οι εκστρατείες στο διαδίκτυο είναι πολύ σημαντικές και είναι περίπου το 70% ε, των συναλλαγών στο διαδίκτυο. Η απάτη βέβαια έχει κόστος. Οποτεδήποτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με μια συναλλαγή κάποιος πρέπει να πληρώσει και ως ε, ρυθμιστές αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε βεβαίως ενδέχεται το κόστος της απάτης να καλύπτεται μέσα στο κόστος που επιβάλλεται στους ε, συναλλασσόμενους αλλά στη τελική ανάλυση όλα αυτά μετακυλίονται στον καταναλωτή στις τιμές καταναλωτή γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί απάτη και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ε, στην δεύτερη αυτή οδηγία ε, η ασφάλεια είναι το βασικότερο στοιχείο για τον ε, νομοθέτη. Βεβαίως υπάρχει ακόμα περιθώριο για εξαιρέσεις ε, και ευελιξία στο κείμενο του επίπεδου 1. Εμείς δεν διαφωνούμε στο να εξετάζονται δυνατότητες για να μπορούν να χορηγούνται δάνεια και με αυτό αυτό, στο πλαίσιο, αυτό το πλαίσιο. Σε γενικές γραμμές εμείς δεν διαφωνούμε με την ανάλυση των κινδύνων, θεωρούμε όμως ότι αυτά λειτουργούν και συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστούν. Άρα δηλαδή σε τελική ανάλυση αυτό που παίζει ρόλο είναι να εξεταστούν ε, οι δανειδοτήσεις ε, και προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο που ήδη σχολιάστηκε ε, σχετικά με την ασφάλεια. Νομίζω ότι και από αυτού ε, τα άρθρα του ε, κειμένου επίπεδου 1 είναι ξεκάθαρα. Η ερμηνεία του άρθρου 67 είναι ότι η διεπαφή μεταξύ των τραπεζών και το ISB είναι ικανοποιητική και θα συνεχιστεί. Το άρθρο 66 της οδηγίας είναι σαφές, διότι απαιτεί από τις τράπεζες να δίνουν όλες τις πληροφορίες ε, για να ξεκινήσει μία πληροφορία και για να εκτελεστεί μία πληρωμή. Να σας εξηγήσω εδώ λιγάκι το εξής. Α, η οδηγία έχει αλλάξει την κατάσταση. Πριν από την οδηγία υπηρεσιών πληρωμών ήμασταν σε μία κατάσταση όπου τα PSP ε, ήμασταν σε μια φάση που υπήρχε μια διεπαφή τραπεζική και τώρα περνάμε σε μια φάση περνάμε σε μια φάση όπου αυτή η οδηγία υπαρθμών 2 θα αλλάξει την κατάσταση. Ε, δεν θα είναι όπως ήταν και είναι σήμερα. Νομίζω οι περισσότερες τράπεζες ε, ε, θα πρέπει να αφομοιώσουν αυτές τις αλλαγές, να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο περιβάλλον και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Μία μεγάλη ανησυχία μας είναι η σταθερότητα και, αυτό, και αυτή η νέα διεπαφή. Ε, ανησυχούμε γιατί αυτή η διεπαφή θα πρέπει να είναι απόλυτα λειτουργική, ε, να λειτουργεί 24 ε, ώρες το 24ωρο, αδιάλειπτα δηλαδή, και να είναι αποτελεσματική η διεπαφή. Γιατί έχουν υπάρξει κάποιες περιπτώσεις που κατέρευσε αυτή η πλατφόρμα. Κατανοούμε βέβαια τις ανησυχίες είναι θεμελιωμένες και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει ε, έξτρα προσπάθεια στο πλαίσιο του ε, provider, του παρόχου και της οδηγίας Πιστεύουμε ότι η λύση θα πρέπει κυρίως ε, να προκύψει από την καλή συνεργασία ανάμεσα στους ε, νέους παρόχους ε, και τους καταξιωμένους, τους παλαιούς γνωστούς παρόχους. Και ελπίζουμε ότι αυτή η τυποποιημένη προσέγγιση που τη βλέπουμε και ως ένα τεχνικό επίπεδο 3, αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν κάποιες ανησυχίες. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, εμείς ε, θέλουμε να βοηθήσουμε να υπάρξει ευελιξία έτσι ώστε κάποιες ανησυχίες που εκφράζονται από τους διάφορους ε, ενδιαφερόμενους να ληφθούν υπόψη. Και όσον αφορά και τη διεπαφή επικοινωνίας, ε, θα πρέπει αυτή πράγματι να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και να σέβεται ε, το γράμμα της οδηγίας της υπαριθμών 2 για την περιπηρεσιών πληρωμών. Επίσης, η πρόταση για τον γεωαποκλεισμό του geo-blocking είναι σημαντική και νομίζω ότι αυτή ε, ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εισηγητής, ο κύριος Σταγιάννη έχει το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ευχαριστήσω και την διαπραγματευτική ομάδα του PSD2, ε, τον κύριο Βέμπερ δηλαδή. Ε, κατά τη διάρκεια των δημοτεύσεων είχαμε πολύ καλή συνεργασία και πολύ καλό κλίμα. Σημαντικό για τα μέτρα επίπεδου 2 και την σωστή του εκπόνηση. Τον περασμένο μήνα, όπω είπε ο κύριο Ένρια, στείλαμε επιστολή προ προς, προς τον Διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, εκφράζοντα ανησυχίε ε, από την πλευρά τη Διαπραγματική Ομάδα για το σχέδιο των τεχνικών πρότυπων. Μεταξύ των ανησυχιών αυτών, η πρόσβαση από τρίτα μέρη και παροχούς Οι αρχικές πληρωμές και οι λογαριασμοί των κατόχων και το TPP. Ε, εδώ συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να μπορούν οι πάροχοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους γνωρίζοντας την εντολή του λογαριασμού ασχέτως άμεσης ή άμεσης πρόσβασης και με συγκεκριμένο πρότυπο παροχή υπηρεσιών. Γι' αυτό ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ειδική διεπαφή. Εκφράσαμε αυτέ τι ανησυχίε στην επιστολή μα. Δεν τι επαναλαμβάνω και δεν επαναλαμβάνω και τα επιχειρήματα. Απλώ να θυμίσω ότι η πολιτική πρόθεση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των δημοκρατήσεων ήταν ευθυμραμισμένη με την πρόταση τη Επιτροπής να ξεκινήσει μια αγορά πληρωμών και να ανοιχτεί τι νέους ε, παρόχους παρόχου ε, με την προσφορά νέων τεχνολογικών λύσεων. Βεβαίω αυτό που είπε ο κ. Ένδια στο λόγο του. Είναι μια καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή και ευχαρίστως να βρούμε μια λύση συμβιβασμού. Όμως πρέπει να ενισχύσουμε τη στρατηγική της οδηγίας για τις ε, πληρωμές. Μπορεί να γίνει αλλαγή στο διαδίκτυο, μπορεί να επιτευχθεί συμβαστική λύση σε τεχνικό επίπεδο. Είμαστε έτοιμοι για συζήτηση, αλλά σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τη στρατηγική και τη φιλοσοφία της οδηγίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Λούντφιξον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλω να πω καταρχάς και να χαιρετήσω την τραπεζική αρχή για τη δουλειά της σε ό,τι αφορά την ε, επεξεργασία της διαδικασίας ταυτοποίησης, η οποία είναι πια ισχυρή. Έτσι έχουμε και καλύτερη συνεργασία υπό την ε, έννοια της ε, Οδηγίε για τις πληρωμέ. Θέλουμε να υπάρχει προστασία των καταναλωτών, προστασία και των παρόχων στο πλαίσιο αυτών των τραπεζικών περιβαλλόντων. Τονίσαμε ότι χρειάζεται ένα κοινό πρότοπο για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και ασφαλή επικοινωνία, προκειμένου να εγγυηθούμε τον πρωταρχικό μα στόχο, την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και την ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής αγοράς. Μια από τις προθε προϋποθέσεις είναι η παροχή πρόσβασης στους ε, παρέχοντες υπηρεσίες πληρωμών. Και να υπάρχουν και πληροφορίες για το λογαριασμό χωρίς να χρειαστεί κάποιο μεμονωμένο μοντέλο. Είτε μιλάμε για άμεση, είτε μιλάμε για έμεση πρόσβαση για τη διάθεση τέτοιων υπηρεσιών. Η υποστήριξη προς την ε, άμεση πρόσβαση προκύπτει από την τελική σκέψη 63, ε, όπως υπόθηκε ήδη. Όμως εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο άρθρο 19 και στα προβλήματα του RTS. Εδώ γίνεται λόγος για μια ειδική υποχρεωτική διαπαθή. Το άρθρο 92.2 ωστόσο αντιφάσκει με αυτήν την ε, διάταξη στη συνολική θεώρηση της οδηγίας. Μιλάμε για βασικές προϋποθέσεις ώστε να έχουν όλη τη δυνατότητα, να έχουν ίσους κανόνες παιχνιδιού και να υπάρχει ουδετερότητα τεχνολογική στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν βλέπουμε να υπάρχουν απόψεις διαφορετικές ως προς τις τεχνικές προδιαγραφέ. Θα πρέπει σε αυτό το επίπεδο να αποσαφινιστεί τι γίνεται με την ταυτοποίηση, και πώς μπορεί να υπάρχει άμεση πρόσβαση. Εφόσον υπάρξει αυτή η ειδική διεπαθή. Σε ό,τι αφορά του παρόχου υπηρεσιών ε, και την πρόσβαση στι πληροφορίε των λογαριασμών, το 66.6 το 66 μάλλον, θα πρέπει να προβλέψει συγκεκριμένε υποχρεώσει στην PST2, ε, ακόμα και αν η ταυτοποίηση συνδυαστεί με την άμεση πρόσβαση. Μέσω ακριβώς της ειδική διαπαφής. Ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει στην εντολή πληρωμής να δείχνει πώς ακριβώς έγινε η ταυτοποίηση. Δηλαδή, να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία όπου ο ε, πληρώνων να λαμβάνει πληροφορίες για τον λογαριασμό. Και αυτό και στο μέλλον, να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες των λογαριασμών, προκειμένου να γίνεται σωστή ταυτοποίηση του ε, πληρώνοντος στο 69 και στο 64-4. Στην περίπτωση του PSD2, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να διασφαλίζουν ότι γίνεται να υπάρξει ταυτοποίηση μέσα τους άμεσης ή έμεσης πρόσβασης. Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην διαπραγματευτική ομάδα ανησυχούν για τις λεπτομέρειες της πρότασης του RTS. Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να επαληθευτούν στις εξαιρέσεις, στην ταυτοποίηση. Το όριο των 10 ευρώ που κατά την άποψή μας είναι πολύ χαμηλό και καλύτερα πολύ μικρό μέρος των συναλλαγών. Ελπίζουμε οι ανησυχίε μας αυτές να ληφθούν υπόψη. Όσα είπαν οι συνάδελφοι της Επιτροπής ΕΚΟΝ πρέπει να ληφθεί υπόψη. και πρέπει τα ζητήματα αυτά να καλυφθούν και στα πλαίσια της οδηγίας PSD2. Με ουδετερότητα, ανταγωνιστικότητα ως προτεραιότητες, με την ανάγκη να βρεθούν λύσεις. Thank you. Um, now for the ECR, Mr. Ευχαριστώ. Από το ECR ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθαν σήμερα να μας παρουσιάσουν τις προτάσεις αυτές. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Για ποιο λόγο αυτό ε, το σχέδιο RTS δεν ε, ακολουθεί ε, την προσέγγιση κινδύνου για την ε, απάτη, όπως είχαμε στο ε, PSD1. Αυτά τα λέει το άρθρο 98 για την ασφάλεια μέσω της υλοποίηση και της έγκρισης ε, των απαιτήσεων που βασίζονται στο κίνδυνο. Εγώ θα έλεγα ότι αν βάλουμε όριο 10 ευρώ ή 50 ευρώ για τις πληρωμές, αυτό δεν είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο. Βάζεις αυθαίρετα ένα ποσό. 25% των απατών στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορά ποσά κάτω των 10 ευρώ. Και υπάρχει καμία ε, δικαιολόγηση ή είναι βολική αριθμή. Γιατί επιλέξατε αυτά τα ποσά. Γιατί εγώ θα σας έλεγα ότι καλύτερα αντιμετωπίζουμε την απάντη να έχουν ένα στόχο η πάροχη υπηρεσιών πληρωμής για να μειωθεί η απάτη κάτω από αυτό το στόχο. Ας πούμε, 10.000 ή 3.000 ή 2.000 και από εκεί και πέρα συζητούμε ποιο είναι το αποδεκτό επίπεδο απάτης ή όχι σε σχέση με αυτό το στόχο. Μου κάνει εντύπωση όμως, αν αντί να βασίζεστε στην ανάλυση με βάση τον κίνδυνο, επιλέγετε ένα ποσό που θεωρείται κατάλληλο. Εγώ δεν δέχομαι ότι αυτή είναι ανάλυση με βάση τον κίνδυνο και θα ήθελα τα σχόλιά σας από αυτού. Και δεύτερον, έχω ένα πρακτικό ερώτημα για τις ανέπαφες συναλλαγές, πώς μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δίκτυα μεταφορό ε, χωρίς να έχει terminal pin. Ε, όταν καμιά φορά χρειάζεται ταυτοποίηση του χρήστη. Όλο και περισσότερο έχουμε ανέπαφες ε, συναλλαγές αντί για το FES εισιτήριο και ως αξιόπιστο σύστημα. Πώς μπορείτε να επιβάλλετε όριο 150 ευρώ ανέπαφων συναλλαγών. Καμιά φορά ε, θα πρέπει να χρειάζεται ασφαλή ταυτοποίηση ε, του χρήστη. Ας πούμε πάει ένας για ψώνια, ε, νέος, και δίνει 149 ευρώ για τα ψώνια και πάει να πάρει αργά το βράδυ το λεωφορείο ή το μετρό και δεν έχει αρκετά λεφτά στην κάρτα του ανέπαφης συναλλαγής και δεν μπορεί να βγάλει εισιτήριο και δεν υπάρχει και ε, σύστημα να το επαναφορτήσει. Τι θα γίνει ας πούμε για ανθρώπους που είναι έξω αργά το βράδυ, έχουν την κάρτα και δεν μπορούν να βάλουν πιν, δεν μπορούν να γεμίσουν την κάρτα τους. Τι είναι αυτά τα αυθαίρετα νούμερα. Thank Ευχαριστώ. Η Σόφι Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τις παρουσιάσεις σας με προσοχή. Ναι, αν ακούσετε τι ανησυχίες έχουν αγερθεί στην επιστολή αυτή τη Επιτροπή, δεν μπορώ να πω ότι έλαβα καμία. ότι καθυσυχάστηκα και καθόλου. Ιδίω με το θέμα της διαπαφή. Διότι πραγματικά έχω την αίσθηση ότι μάλλον η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό με τόσο ενθουσιασμό όπως μια γαλοπούλα που διζητήθηκε ζητήθηκε να ετοιμάσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Έχω την εντύπωση και αυτή την αίσθηση έχουμε εκφράσει και στην επιστολή ότι χρησιμοποιείται το θέμα της ασφαλείας και προστασίας δεδομένων προκειμένου ο ανταγωνισμός να μείνει εκτός. Και ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει στην πράξη. Αυτό κάνουν οι τράπεζες σήμερα. Χρησιμοποιούν αυτές τις δικαιολογίες για να κρατήσουν εκτός τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής και παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες οι ίδιες. Βρίσκω ότι είναι κατάχρηση της θέσης των τραπεζών αυτή. Και δεν είμαι καθόλου πεπισμένη από την απάντησή σας και θεωρώ ότι η τελική μορφή των τεχνικών προτύπων θα πρέπει να δίνει μια απάντηση στις ανησυχίες που εκφράσαμε ώστε πραγματικά αληθινά ο ανταγωνισμός και η καινοτομία να ε, υπάρξουν και όχι απλώς να είναι εργαλεία ώστε ύπουλα να μπλοκάρουμε τις αλλαγές και την καινοτομία. Αυτό το παιχνίδι το παίζουν ε, αρκετό καιρό οι τράπεζες. Χρησιμοποιούν το πρόσχημα των ε, προτύπων για να αφήνουν εκτός αγοράς τους ε, νέους που θέλουν να μπουν εκεί και να παρακρατούν πληροφορίες. Ενώ πολύ γρήγορα αναπτύσσουν τις δικές τους εσωτερικές υπηρεσίες για να ανταγωνίζονται με τους υπόλοιπους. Αυτό κάνουν με το μοντέλο τους και χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών, των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών, ως εργαλείο. Πραγματικά το βρίσκω αρκετά αξιόμεμπτο αυτό και Ελπίζω ότι τα πρότυπα που θα εκπονηθούν να είναι πρότυπα που θα επιτρέπουν πραγματικά έναν υγιή ανταγωνισμό, να υπάρξει πραγματική καινοτομία και όχι απλώ να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα ενό μέρους των ε, επιχειρήσεων του χώρου αυτού, αλλά να υπάρξει πραγματικό άνοιγμα τη αγορά. Ευχαριστούμε. Ο Ματ Κάθι Δεν είναι εδώ. Ο. Και εδώ για τους ε, πρασίνους ο Σβέν Κίγκολτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, επιτρέψτε μου ε, με την ε, συμμετοχή μας στις ακροάσεις αυτές, αφού απορρίψαμε τα πρότυπα BEPS, Πραγματικά χαίρομαι που εδώ τουλάχιστον υπήρξαν κάποιες αλλαγές στη σύνθεση. Είναι τα έδρανα γεμάτα και έχουμε πάρα πολλούς ε, φορείς και θεσμούς που εκπροσωπούνται ταυτόχρονα. EBA, ACT και ούτω καθεξής. Έχει αλλάξει κάπως η εικόνα λοιπόν. Θετικό αυτό. Θετική εξωτερική επιρροή. Έχουν ακουστεί πολλά επιχειρήματα και δεν θέλω να τα επαναλάβω. Θέλω απλώς να πω το εξή. Πριν την ανταλλαγή μας, πριν τη συζήτηση δηλαδή, σημαντικό είναι να δούμε πόση άσκηση πίεση θα υπάρξει, πόσο λόμπινγκ. Οι τράπεζε ανησυχούν πολύ για την προστασία των δεδομένων. Πάντοτε όταν μου τίθεται τέτοιε ερωτήσει, αρχίζω και γίνομαι καχύποπτο. Από την άλλη, νομίζω ότι οι αρχές ανταγωνισμού ανησύχησαν πραγματικά για την πρόταση του RTS. Και η αρχή της Γερμανίας κατά τον καρτέλ μου λέει ότι αυτός ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να υπάρξει ε, για τον κλάδο αυτό και να μην υπάρξουν αδικαιολόγητα περιθώρια. Θα μας ενδιαφέρει πολύ να μάθουμε τι άποψη έχει σχετικά η Γενική Διεύθυνση ΚΟΜΠ. Και από εκεί να είχαμε καμιά απάντηση. Όμως η δική μου εντύπωση είναι ότι το κείμενο έχει επειδή δεν προβλέπει και πολλά για την έμεση πρόσβαση, δεν συνάδει με το ένα, με το επίπεδο ένα. Και εφόσον υπάρχουν ανησυχίε περί ασφαλεία, βεβαίω θα μπορούσαν να καλυφθούν με το να προβλεφθεί υποχρέωση, ώστε να απαιτείται από τι τράπεζε και ίσω και από τα τρίτα μέρη να κλειδώνουν την πρόσβαση που ήδη έχει λάβει χώρα, κάτι που τεχνικώ είναι εφικτό, παρά να κόβουν την άμεση πρόσβαση, την απευθεία πρόσβαση. Ή να επιτρέπουν τι τράπεζε να παρεμποδίζουν τα τρίτα μέρη από την απέτηση την απέτηση και από τις δύο πλευρές τις τράπεζες και τους παρόχους ως τρίτα μέρη να κλειδώνουν την πρόσβαση στα δεδομένα. Έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη επίπεδο ασφαλείας. Χωρί να περιορίζουμε όσο προβλέπει και το κείμενο του επίπεδου 1, περισσότερο ανταγωνισμό και περισσότερη παρουσία φορέων, πολυφωνία. Μα ενδιαφέρει κυρίω όμω η απάντησή σα για το τι λένε οι αρχές ανταγωνισμού και ποιε είναι οι απόψει τη γενική Διεύθυνσης ΚΟΜΠ. Ευχαριστούμε πολύ. Μάρκο δεν είναι παρόν. Κύριε Πάλτς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι κανένα δεν θα πρέπει να εκπλήξει το γεγονός ότι η δική μας πρόθεση ως ΕΚΟΝ σήμερα είναι να υπενθυμίσουμε την ε, απόφαση αρχής ε, των συνομοθετών. Δεν πρόκειται μόνο για την τεχνική εργασία, αλλά και για βασικά θέματα της πρόσβασης στην αγορά και του ανταγωνισμού. Αυτή η οδηγία υπηρεσιών πληρωμών υπαριθμών 2 καθορίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση στον ανταγωνισμό. Το ξέρει η Κομισιόν, το ξέρει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και η ΕΚΤ. Κατά την άποψή μου λοιπόν ε, εδώ δεν θα τσακωθούμε για το κατά πόσον οι αρχές αυτές ε, θα πρέπει να αναφέρονται σε οδηγήσεις σε σκεπτικό. Το θέμα είναι ότι ήταν πάντα ένα κομμάτι της ε, πολιτικής ολοκλήρωσης. Και ως Κοινοβούλιο εμείς πάντα θα μεριμνούμε στο να αναζητείτε μια τεχνική λύση ακριβώς όπως είναι η στόχη της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ουδετερότητας ισότητα στον ανταγωνισμό να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι γιατί με τον τρόπο αυτό ε, θα μπορούμε να ε, βοηθήσουμε τον καταναλωτή να υποφεληθεί από αυτές τις ανέπαφες ε, πληρωμές. Η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι ήδη τώρα σε κράτη-μέλη υπήρξαν έρευνες που κατέληξαν στο ότι πρέπει να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Η δική σας η εργασία πώς μπορεί να προωθεί στον ανταγωνισμό. Και μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Θα αποκλίνεται από τις ε, αποφάσεις της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Εποπτικής Αρχής αν, λάβετε, δείτε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις σας. Υπερβάνσου Σπέρες, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι συζητήσει αυτές έχουν ξεκινήσει από καιρό. Ούτε που θυμάμαι πότε συζητήσαμε πρώτη φορά το πρώτο κείμενο. Και τα λόμπι δεν έχουν αλλάξει η αναδιανομή, οι τράπεζες, η παροχή και οι υπόλοιποι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει εδώ είναι η προστασία των καταναλωτών ε, με την πραγματική της έννοια. Και επίσης οι τράπεζες θα κάνουν και τη δουλειά τους. Δεν είμαι λομπίστας υπέρ των τραπεζών. Αλλά πρέπει να υπάρχει η εποπτεία, η διανοητική ικανότητα, και αφήνω τα καλύτερα. Δουλειά των τραπεζών είναι να δανείζουν χρήμα. Αλλά βλέπουμε τις τράπεζες να έχουν ε, μαζέψει χρήμα και να προσπαθούν να μεταλλευόμενε την τεχνολογία να μπουν σε ένα νέο κλάδο. Τι υπερεταζόμαστε σήμερα τις τράπεζες, τα, αύριο τα σούπερ μάρκετ και προχθές τους νέους παρόχους υπηρεσιών. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα στο θέμα της ασφάλειας ε, των συνελλαγών της υπηρεσίας που παρέχεται πλέον σε αυτούς τους καταναλωτές, πρέπει ως νομοθέτες να είμαστε λιγάκι συνεπείς. Και θα προσθέσω ένα στοιχείο που καθόλου δεν αναφέρθηκε σήμερα. Όταν βλέπω το τι υποθέσει απάτη έχουν τον πεστεί την Επιτροπή, αρχίζω και ανησυχώ. Στην ομάδα των Σοσιαλιστών τη προάλλε, η ο σύντροφός μας Λόπες Αγγιλάρ μας έλεγε ότι ο πρώην συνάδελφος Μπορέλ έπεσε θύμα, α, έτσι, μίας ε, υπεξαίρεσης από τον τραπεζικό του λογαριασμό χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτό λοιπόν είναι το πνεύμα του νομοθέτη στο επίπεδο 1 όταν προασπίζεται τα στοιχεία ασφάλειας θα πρέπει να είναι και αρκετά σοβαρά. Η ειδική διεπαφή δεν είναι για να εμποδιστεί η καινοτομία, οι νέοι πάροχοι ή να διευκολύνεται μόνο ο καταναλωτής. Ανασυχούμε με το διπλό κλικ επαλήθευσης όταν αγοράζει κανείς το ίντερνετ. Ε, τι λέτε, το κάναμε όλοι. Το να πάρει κανεί ένα γραπτό μήνυμα για να επιβεβαιώσουμε τον κωδικό αυτό την ταυτότητα μέσω τη τράπεζα δεν μου φαίνεται και φοβερό όταν ξέρουμε τι επίπεδο απάτη υπάρχει στο ίντερνετ. Και να προσθέσω και ένα στοιχείο που δεν αναφέρθηκε καθόλου και που γνωρίζω ότι μας απασχολεί στη Γαλλία όπως και σε άλλα κείμενα είναι αυτό της διαπαθής. Δεν θέλω να διευκολύνουμε τόσο πολύ τη διαπαθή που να μην ελέγχουμε πια τίποτα. Καταλαβαίνω κάποιες από τις ανησυχίε που εδώ εγέρθησαν Όμω και πάλι να ζητήσω από την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή τι απάντηση δίνουν σε αυτό το κίνδυνο μη εποπτεία και ασφάλεια των πληρωμών που οπωσδήποτε ήταν ένα από του στόχου του πρώτου επίπεδου. Ευχαριστούμε ο κύριος Βέπερ. Äh, σας ευχαριστώ πολύ. Είχα την τιμή να προεδρεύω ε, στον τριμερή διάλογο και έχω υπογράψει και αυτή την επιστολή που αναφέρατε. Να σας υπενθυμίσω μόνο ότι σε αυτή την δεύτερη οδηγία δεν μας ε, ενδιαφέρει ε, να απορρίψουμε κάποιες δυνατότητες από την αγορά, αλλά του αντίον να ανοίξουμε τον δρόμο. Και αυτό είναι προς όφελος του καταναλωτή, είναι υπέρ της προστασίας του καταναλωτή και γι' αυτό το άρθρο 98.2α ε, αναφέρθηκε ήδη. Εκεί αναφέρεται ότι ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, αιτήματα που να βασίζονται σε υπάρχοντες κινδύνους εγώ αυτό όμως δεν βλέπω εσείς να το αναφέρετε. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας καλός ε, συμβασμός ανάμεσα στα συμφέροντα των τραπεζών ε, και στα συμφέροντα των νέων παρόχων. Κατά την άποψή μου κανείς δεν έχει απόλυτα δίκιο, αλλά τελικά καθήκον της ε, πολιτικής είναι να βρίσκει μια εξισορροπημένη πρόταση και η κριτική την οποία θέλαμε εμείς να εκφράσουμε με την επιστολή μετά από συζήτηση με τη διαπραγματευτική ομάδα δεν ήταν η ισορροπία που έπρεπε να αναζητηθεί. Ας πούμε, ε, εισιτήριο κινηματογράφου 10 ευρώ, κανείς δεν πάει στον κινηματογράφο για 10 ευρώ. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς ε, να τα ρυθμίζει όλα μέσα από τους παρόχους. Και εάν έχω καταγραφεί και έχω δώσει κάποιες πληροφορίες, αντιμετωπίζω τελείως διαφορετικό κίνδυνο από το να είμαι καινούριο σε κάποια πλατφόρμα. Αυτό το κίνδυνο πρέπει κανείς να τον αξιολογήσει διαφορετικά, γιατί υπάρχουν ήδη κάποια στοιχεία. Αν πρόκειται για μία γνωστή συσκευή, αυτό το ξέρουμε και με την ηλεκτρονική αλλογραφία. Βλέπουμε ότι προσπαθεί κάποιος ε, να μπει στο ε, λογαριασμό σας μέσα από μία ε, συσκευή που δεν είναι γνωστή. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα πάρα πολλές δυνατότητες και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν θέλω και εγώ να ερωτήσω αυτό το άρθρο 98.2α πώς μπορείτε να του δώσετε σάρκα και οστά γιατί απλά και μόνο οι ανώτατες τιμές για μένα δεν βασίζονται στην αξιολόγηση κινδύνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτό το θέμα των οριακών τιμών συμφωνώ. Για το άλλο θέμα της διαπαφής προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζεται μια ισόρροπη προσέγγιση να λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία της νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 66.3 ε, εδάφιο που ζητεί ε, ότι κάθε φορά που θα υπάρχει ε, συναλλαγή πάνω από ένα ποσό να υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς ταυτοποίησης του πελάτη του χρήστη. Εγώ δεν το βρίσκω πάρα πολύ αντιφατικό αυτό με τα όσα λέγει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Είναι πολλές ερωτήσεις για σας λοιπόν. Δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές είναι όντως ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικές και στις υπόλοιπες CBA. από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ανάλυση βάση κινδύνου ή το TRA που ανέφεραν δύο-τρεις ευρωβουλευτές. Εγώ δεν θέλω να μπω τώρα σε μια μακρά ε, και κουραστική νομική ε, αντιπαράθεση. Αλλά το άρθρο 98 του PSD2 οδηγίας θα πρέπει να αναγνωστεί σωστά. Προβλέπει εξαιρέσεις ε, με βάση διάφορα κριτήρια που είναι πολλά. Πρώτον είναι το επίπεδο του κινδύνου της υπηρεσίας, το δεύτερο είναι το ποσό της συναλλαγής και το τρίτο είναι ο διάβλος πληρωμής που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση αυτής. Άρα δεν ανοίγει διάπλατα τη θύρα για το RPA, αλλά το RPA που είναι ανάλυση με βάση το κίνδυνο, δηλαδή risk-based analysis, Υπάρχει χώρο δεν είναι αντιφατικό, επαναλαμβάνω. Και θα μπορούσε αυτό να είναι συμπληρωματικό, αλλά όχι πλήρες υποκατάστατο. Θα το ξαναδούμε όμως αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, θα το ξανακοιτάξουμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μπορεί να έχουμε και κάποια μεγαλύτερη ευελιξία για τα κατόφλια ήταν οι ανώτατες ε, τιμές τα ποσά. Στο σχέδιο του Αυγούστου τη CBA ακριβώς αυτός ήταν ο στόχος. Ήταν ένα προσχέδιο για διαβούλευση και περίμεναν τις απαντήσεις των διαφόρων ε, ενεχομένων και ενδιαφερομένων. Και είναι ε, πιθανότατο το τελικό σχέδιο να είναι κάπως διαφορετικό. Για τα σχόλια που έκανε η κυρία Εντβέλτ και άλλοι ευρωβουλευτές το είπα στην αρχική μου τοποθέτηση και βέβαια ο ανταγωνισμός είναι ένας από τους βασικούς στόχους ε, της οδηγίας ε, για τις υπηρεσίες πληρωμών PSD2. Αλλά υπάρχουν και άλλοι στόχοι στην ίδια νομοθεσία. Ε, άλλο στόχο είναι η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια. Και η κυρία Περβάν ε, Μπερέ πολύ σωστά θύμισε το θέμα της προστασίας των καταναλωτών και την ευγνωμονώ γι' αυτό. Εδώ μάλλον καλούμαστε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο ε, πολύ συγκεκριμένα μεταξύ των τριών αυτών στόχων. Για να κάνω μια σύγκριση πριν από λίγα χρόνια, ότι όταν βάλαμε το διπλό chip και πιν ε, ήταν σχεδόν επανάσταση. Όπως γίνεται τώρα ε, με την αναγνώριση για τις επιγραμμικές προμές και χρειάστηκε χρόνος για να ε, προσαρμοστούν όλοι οι χρήστες και οι ενδιαφερόμενοι και οι πελάτες και οι πάροχοι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά κάποιες από τις ανησυχίες που αναφέρθηκαν και εδώ. Εργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με το κείμενο του Αυγούστου, αλλά θα πρέπει να βασιστούμε το βασικό στόχο ε, της οδηγίας για τις πληρωμές ε, και ως προς το γράμμα και ως προς το πνεύμα, γιατί κανείς δεν έχει την πρόθεση να το ξανανοίξει αυτό, ή να το αμφισβητήσει. Ποιος ε, ακολουθεί τώρα, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους εκείνους που μίλησαν με κίνδυνο να ε, παραλάβω κάποια πράγματα που είπε ήδη ο Λιβιέ. Θέλω να τονίσω πάρα πολύ ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, πιστέψτε με, για να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε όλους τους στόχους ε, του κειμένου της πρώτης οδηγίας. Και δεύτερη οδηγία προσπαθεί να ανοίξει την αγορά ε, σε νέους συμμετέχοντες για το μέλλον και να κάνει κι άλλο ένα άλμα αυξάνοντας την ασφάλεια. Δηλαδή και τα δύο αυτά άλματα θα πρέπει να συμβαδίζουν και να είναι τελικά υπέρ του καταναλωτή και του πελάτη. Εγώ αντικρούω το επιχείρημα στεναρά που λέει ότι έχουμε έρθει εδώ για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων. EBA λεγόμαστε κι εμείς, αλλά είμαστε Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, δεν είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών που έχει τα ίδια αρχικά μαζί μας. Αυτό προσπαθούμε και το είπα και στην αρχή και το τόνισα, ακριβώς να δούμε ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε. Έχουμε διάφορους ενεχομένους ε, συμμετέχοντες που απαντούν ε, για να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Τη βρήκαμε. Ε, είναι έγγραφο Είμαστε πρόθυμοι να δούμε τα διάφορα σχόλια και να τα συζητήσουμε. Και η διαπραγματευτική μας ομάδα και η δική σας στην επιστολή σας τα αναφέρει αυτά. Βεβαίω καλωσορίζουμε αυτή την ε, ευκαιρία για το διάλογο. Τώρα, στις λεπτομέρειες των ερωτήσεων για τις οριακές τιμές και τα ποσά και γιατί δεν έχουμε μια ανάλυση και εξαιρέσει με βάση τον κίνδυνο. Μα ξαναδείτε το άρθρο στο σχέδιο του RTS των ε, τεχνικών ε, κανονιστικών προτύπων. Αναφέρονται αυτά, ας πούμε, η δυνατότητα να ε, βασίζεται σε κάποια δεδομένα ένας πελάτης που έχει τακτικές ε, συναλλαγές με κάποιο πάροχο. Ο Λιβιέ αναφέρθηκε και στην εντολή που είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς βασιζόμαστε στις στατιστικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να δούμε και τα διάφορα ποσά που συνδέονται με κίνδυνο και με απάτη ε, στις διάφορες συναλλαγές. Όπως είπα και στην αρχή, Ερώτηση για τη διαβούλευση είναι. Θεωρείτε σωστά αυτά τα ανώτατα όρια ή τα ποσά ε, ή τα κατώτατα. 10 ευρώ ας πούμε για ε, πληρωμές εξ αποστάσεως μπορεί να είναι πολύ χαμηλό ποσό. Δεν ξέρω, θα το συζητάμε. Γενικά θα έλεγα ότι προσπαθούμε να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες και να απαντήσουμε ε, στα ερωτήματα, στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου, αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τους στόχους που είναι ε, και στόχου ανταγωνισμού και ανοίγματο της αγοράς αλλά και προστασία του πελάτη, στο PSD2, την οδηγία για τις υπηρεσίες ε, πληρωμών. Ε, εμάς μας έχουν αναθέσει να παράγουμε τεχνικές προδιαγραφές και μέσα σε ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει το, ε, η οδηγία για το πρώτο κείμενο. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω μόνο δύο πράγματα να επισημάνω. Σύμφωνο απόλυτα με τον Αντρέα που είπε ότι δεν είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των τραπεζών. Η ΕΚΤ ποτέ δεν ε, έλαβε μια θέση που να προστατεύει τα συμφέροντα των τραπεζών, αλλά ούτε και των μη τραπεζών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο σκέλη, ο πραγματικός ανταγωνισμός. Για τη τελική ανάλυση, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να ε, δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής και ευρωπαϊκής αγοράς ε, για την ε, ε, ε, την παροχή πλησιών ένα πληρωμών. Ε, δηλαδή, να υπάρχουν πολλά TPPs που να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και όλοι να βρίσκουν ένα εύκολο τρόπο ε, για να υπάρχει πρόσβαση στους ενωσιακούς λογαριασμούς οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Άρα δηλαδή η κοινή διαπαυτή είναι ένα στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση γιατί αλλιώς οι TPP θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες να δουλέψουν σε πέντε διαφορετικές διεπαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος της κοινή διεπαφή, δηλαδή να τεθούν τα θεμέλια για μια ανταγωνιστική αγορά. Ε, Ω εκ τούτου, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κανένα ανταγωνισμός ανάμεσα σε κοινό ή ε, τυποποιημένη, κοινή τυποποιημένη διεπαφή. Το επόμενο. Κατά την άποψή μου εκφράστηκε μια ανησυχία που είναι σοβαρή και θα πρέπει πράγματι να λαμβάνεται υπόψη. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε εξαιρέσεις αλλά όχι με τον τρόπο που θα σημαίνει ότι ε, μειώνεται η απέτηση για μεγαλύτερη ταυτοποίηση. Παραδείγματο χάρη η ιδέα ότι θα πρέπει οι εξαιρέσει από την ανάλυση κινδύνου να βασίζονται σε κάτι που οδηγούν αυτήν την ανάλυση να φτάνει σε αποτέλεσμα που θα είναι ε, εξίσου σημαντικό και σωστό όπως και η εξουσιοδότηση αυτό ε, γιατί να μην το εξετάσουμε. Ευχαριστούμε, εισηγητή. Σας ευχαριστώ εν είδη συμπεράσματο. Να προτείνω μια τεχνική συνάντηση για να βρούμε μια λύση. Πρέπει να γίνει μια τέτοια συνάντηση και είμαστε έτοιμοι για συμβασμό. Το σημαντικό δηλαδή είναι να τονίσουμε ότι πνεύμα της οδηγίας αυτής είναι να ανοίξει οδηγία πληρωμών σε νέους φορείς και σε τεχνολογικές λύσεις που να είναι καινοτόμες, νέες. Δεν είμαστε κατά των τραπεζών, να θέλουμε μια λύση εδώ, όλοι θέλουμε την καλύτερη. Πραγματικά προτείνω μια τεχνική συνάντηση αμέσως για να βρεθεί μια συμφωνία. Βεβαίως, ήθιστε να υπάρχει περαιτέρω συζήτηση και προβλέπετε να συζητήσετε με την ε, ΕΤΑ και την ε, Επιτροπή. Είναι εφικτό λοιπόν αυτό. Πέραν τη συζήτηση εντό Κοινοβουλίου, διότι με το πνεύμα συμφωνούμε όλοι. Το όλο ερώτημα είναι προσωπικό τουλάχιστον, εάν η διαπαφή θα είναι εργαλείο για να πετύχουμε τη μεγαλύτερη προστασία. Εκεί μπορεί να υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Τη συζήτηση λοιπόν αυτή μπορούν να την συζητήσουμε και είναι σκοπιμότατο αυτό που προτάθηκε περί τεχνικής συνάντησης. Ο κύριος Φόξ, παρατηρώ ότι κανείς από τους ειδικού μας σήμερα δεν απάντησε στην ερώτησή μου για τον νεαρό που ξόδευε 149 στο σούπερ μάρκετ και μετά πάει να πάρει το τρένο ή το λεωφορείο και δεν μπορεί να πάει σπίτι του. Ίσως κάποιος με όλες αυτές τις προτενέμενες λύσεις του όσα ακούσαμε να μας τα απαντήσει, διότι αν δεν υπάρχει απάντηση υπάρχει και ένα κατάφορο πρόβλημα για τους καταναλωτές. Ναι. Ακούω με θετικό αυτή όσα υπόθηκαν. για το ότι χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες. Αυτό που κι εσείς παρατηρήσετε είναι πολύ σκόπιμο. Δεν θα πω για τη δική μου περίπτωση εξαπάτησης. Μου συνέβη και εμένα πρόσφατα και υπερβάνης μας θύμισε μια άλλη. Νομίζω το Κοινοβούλιο θα παραμένει σε επαφή με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συνεδρία.